Okay, good morning. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους ε, ευρωβουλευτές που ήρθαν σήμερα το πρωί. Καταρχήν να σας ε, υποβάλω προς έγκριση κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν το σημείο 7 της αρχικής ε, διάταξης, συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ, θα είναι το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης μετά τις ανακοινώσεις. Επίσης, το, το σημείο προστασία των προσωπικών δεδομένων από τους ε, ε οργανισμούς ε, γραφεία και ούτω καθεξής και την ελεύθερη κυκλοφορία, αυτό θα συζητηθεί γύρω στις 9 και 20. Θα ακολουθήσει το σημείο 6, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας για τους ε, συμπληρωματικούς κανόνες ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική στήριξη για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις ε, ως τμήμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020. Το σημείο αυτό θα συζητηθεί γύρω στις 10 παρα 10 μετά θα επανέλθουμε στο σημείο 4 για την αμοιβαία αναγνώριση των ενταλμάτων δέσμευσης και δίμευσης. Αυτό θα συζητηθεί γύρω στις 10. Αυτές είναι οι αλλαγές που προτείνω στην ημερήσια διάταξη και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις παρακαλώ να την εγκρίνουμε με τις αλλαγές αυτές. Σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, δυστυχώς σήμερα δεν θα έχουμε διερμηνία στα κρατικά, λετωνικά και γοεδελικά. Ούτε το απόγευμα δυστυχώ, δεν θα έχουμε δανέζικα, κροατικά και εγωεδελικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών, ορισμό εισηγητών. Ο κύριος Έγκελ από το ΕΛΚ ορίστηκε εισηγητή για την ετήσια έκθεση που αφορά την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για το 2016. Η κυρία post από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες θα αναλάβει την έκθεση πρωτοβουλία για τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την, ε, την, ένταξη, την κοινωνική ένταξη στο Ρωμά και την καταπολέμηση της, του αντιαθηγανισμού. Επίσης, ο κύριος Μπόνι έχει οριστεί εισηγητή τη γνωμοδότηση ε, για την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου για τα θέματα copyright στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Μπορούμε να εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών δυνάμει του άρθρου 205. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Οπότε περνάμε στις κατεξουδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Στις 24 Μαρτίου 2017 η Επίτροπος Γιώροβα έστειλε επιστολή στους Προέδρους των Επιτροπών Οικονομικών Πολιτικών Ελευθεριών και Επιτροπής του Παναμά μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφέρει αντιρρήσει στην κατεξουδότηση πράξη τη 24η Νοεμβρίου του 2016 που συμπληρώνει την οδηγία, την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε μια νέα κατεξουδότηση πράξη ε, με τον αναθεωρημένο κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου. Και μάλιστα το έχουμε λάβει στο Λιμπεντία και στο δελτίο το ενημερωτικό την περασμένη ε, Παρασκευή. Η νέα κατεξοδότηση πράξη αφαιρεί τη Γουιάννα από τον κατάλογο ε, αυτών των ε, χωρών υψηλού κινδύνου και συμπεριέλαβε την Αιθιοπία. Έχουμε ένα μήνα για να εκφέρουμε αντιρρήσει. Οι ΛΥΜΠΕ και οι ΕΚΟΝ έχουν κοινέ αρμοδιότητε δυνάμει του άρθρου 55. Η εσωτερική προθεσμία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για υποβολή αντιρρήσεων με την μορφή σχεδίου ψηφίσματο. Η προθεσμία αυτή λήγει στι 6 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Παρόμοια προθεσμία έχει θεσπίσει και η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σε περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις, παρακαλώ στείλτε την, το αιτιολογημένο σα αίτημα ψηφίσματο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Πρόεδρο και την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πριν την εκπνοή της προθεσμίας. Έχουμε και έγκριση κάποιων πρακτικών από τον Ιανουάριο φέτος, από τον Νοέμβριο του 2016, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Φεβρουάριο του 2016 και αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε στα κυρίω θέματα. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της τροποποιημένης, Πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Ντίας Δεμέρα για το σχέδιο συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγική συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και του Βασιλείου της Δανημαρκίας. Κύριε Ντεμέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω πρώτα μια σύντομη δήλωση που αφορά ε, τον άνθρωπο, τον Άγα Γιώρες που κάθεται εκ δεξιών σας γιατί από ό,τι ξέρω σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα ε, του κυρίου Γιώρενς στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας μου, αλλά και προσωπικά, να κάνω μια δήλωση. Πρόκειται για έναν κορυφαίο επαγγελματία, ε, εξαιρετικό άνθρωπο, με ιόβια υπομονή, πολύ επιμελή και εργατικό άνθρωπο. Και θα είναι τεράστια πόλια για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Είχα την τιμή και το προνόμιο να συνεργαστώ μαζί του σε πολλά ε, νομοθετικά θέματα και πραγματικά έμαθα πολλά από τη συνεργασία μας. Πολύ καλός φίλος. Και ας περάσουμε τώρα στο νομοθετικό μας σχέδιο. Θα παραλείψω όσα ήδη γνωρίζετε και θα έρθω στο ψαχνό. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Συνεργασίας ε, Επιχειρησιακής και Στρατηγικής με τη Δανία. Έχει εξαιρετικό χαρακτήρα αυτή η συμφωνία, που δεν είδαν ε, ε, θα αντιμετωπιστεί η Δανία ως πλήρες μέλος της Ευρωπόλ. Και μάλιστα παρακολούθησα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η γνώμη μας, όπως είχε παρουσιαστεί στην προηγούμενη έκθεση, ελήφθη υπόψη σε αυτό το σχέδιο και ε, εισακούστηκαν οι παρατηρήσεις μας και οι όροι που θέσαμε. Δηλαδή, η συμφωνία να εξαρτηθεί από την παραμονή της Δανίας στο χώρο Σέγγεν και να συναντευτεί με την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως και να ενσωματώσει στη Δανέζικη ε, νομολογία την τροπολογία 2016-680 για την προστασία των δεδομένων και μάλιστα πριν την 1η Πέμπτου 2017 και τη Συμφωνία της Δανίας ε, να εφαρμόσει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να αναγνωρίσει την ε, αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Νομίζω ότι ο Γιάννα Αλμπρέχτ ε, θα μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις διατάξεις αυτές. Και μάλιστα ε, έχουμε στο αιτιολογικό όλα αυτά τα θέματα 27 κεφάλαια, 27 άρθρα, 7 κεφάλαια και ε, τρία παραρτήματα συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία αυτή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τη δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης του Συμβουλίου η Ευρωπόλ ε, μπορεί να συνάψει τη Συμφωνία Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της Ευρωπόλ. Και δυνάμει του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ε, τίθεται συζητή την ημέρα της κοινοποίησης. Στο χρονοδιάγραμμα που προτείνω εγώ, πέραν τη σημερινή συζήτηση, έχουμε 5 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, εξέταση των τροπολογιών 11 και 12 Απριλίου, Τρίτη ή Τετάρτη, ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στις 27 Απριλίου, ημέρα η θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή στη Μήνη Ολομέλεια. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δίας Δεμέρα και καταρχήν σας ευχαριστούμε για τα πολύ ευγενικά σας λόγια με τα οποία αναγνωρίσατε το αξιόλογο και πολύτιμο έργο της γραμματείας και των υπαλλήλων μας ε, που πραγματικά η συνεργασία μας μαζί τους είναι ανεκτήμητης αξίας. Ευχαριστώ. Κύριος Πίτερσον. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω δανέζικα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για μία ακόμα φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την ε, μεγάλη δέσμευση την οποία ε, έδειξε και την απόλυτα επικοδομητική διάθεση για να βρεθεί συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της Ευρωπόλ. Αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και να το πούμε καθαρά. Επίσης, πρέπει να πω ότι ε, σε σχέση με συμφωνίες αυτού του είδους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια στιγμή η Επιτροπή θα κάνει αναθεώρηση της συμφωνίας, πότε θα προχωρήσει σε εξέταση για να δει εάν πραγματικά λειτουργεί ή όχι η συμφωνία. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και εδώ σε εμά. Εμείς λοιπόν θα υποβάλλουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά εξ αρχής πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε και η προσέγγιση είναι πολύ θετική θετική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία ε, Ζίπχολ έχει το λόγο. Ζίπελ. Ε, στον εαυτό μου δηλαδή. Ε, μπερδεύτηκα λίγο γιατί ούτε στο κείμενο της Κομισιόν ούτε στο κείμενο του συναδέλφου μέρα βλέπουμε να υπάρχει σαφής ημερομηνία και προθεσμία, ε, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή ε, στο τέλος διαδικασίας να έχουμε ε, μια διεθνή συμφωνία γιατί εγώ διαβάζω στο αγγλικό κείμενο ότι η Κομισιόν ενδεχομένως, μει ενδεχομένως να έρθει σε συμφωνία νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί επίσης 5η Απριλίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και παρακαλώ πολύ να υποβάλλετε μόνο στα αγγλικά τις τροπολογίες σας. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Μίτσι, θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα τα οποία είδα ή τα οποία είπα ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Από πλευράς της Κομισιόνη είναι σημαντικό αυτό το σχέδιο συμφωνίας να, να σέβεται ε, την θεσμική ισορροπία καθώς επίσης ε, και τις προϋποθέσεις οι οποίες είχαν αναφερθεί στην κοινή δήλωση του των Προέδρων ε, Γιούνκερ και Τούσκο και του Πρωθυπουργού κ. Ράσμουσεν όπως ε, είπε και ο κύριος ε, Ντεμέρα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να γίνονται σεβαστές ε, πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν αναγνώρισε ότι το προσχέδιο λαμβάνει υπόψη και τα σχόλια της κοινή εποπτικής αρχής της αρχής επίσης εποπτείας της Europol αυτό το θεωρούμε πολύ θετικό βήμα όσον αφορά τα σχόλια τα οποία ε, υπευλήθησαν από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή σας κυρίως όσον αφορά την ε, λήξη της συμφωνίας να σας πω ότι η ημερομηνία της 25ης ε, ε, ανεθεωρήθη έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη ε, και τα σχόλια του Κοινοβουλίου και στο άρθρο 25 προβλέπεται μία ισχυρή ρήτρα αξιολόγησης και αναθεώρηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της συμφωνίας ε, και ε, της συμμόρφωσης ε, της Δανίας όσον αφορά όλους τους κανόνες μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2020. Η έκθεση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα γίνει λοιπόν συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και ανάλογα με το, την έκβαση της αξιολόγησης αυτής, ενδεχομένως θα υπάρξει μία σύσταση από πλευράς της Κομισιόν προς το Συμβούλιο, ζητώντας από το Συμβούλιο να επιτρέψει ε, την ε, εκκίνηση ε, συμφωνιών, διαπραγματεύσεων, συγγνώμη, βάσει του άρθρου 118 της Συνθήκης Λειτουργίας της Λισαβόνας η ενεργοποίηση της ε, ρήτρας ε, που αναθεωρήθηκε, όπως σας είπα, στη διάρκεια της συζήτησης, ε, βάσει αυτής της αναθεώρησης η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει καλύψει τα θέματα της αξιολόγησης, δηλαδή προβλέπει μια ισχυρή αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, δεν αμφιβάλλουμε ότι θα λειτουργήσει καλά η συμφωνία. Πρόκειται κυρίως ε, για πολιτικό ε, ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει η Δανία για το κατά πόσο θέλει να συνεχίσει στην οδό αυτή. Κύριε Ντίας Δεμέρε, θέλετε να ξαναμιλήσετε. Παρακαλώ. Δεν έχω τίποτα πολύ συγκλονιστικό να πω, αλλά ε, θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Μόρτιν Πέρτασεν ε, για αυτά που είπε και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον ε, τις τροπολογίες του, οι οποίες ελπίζω να μην είναι δύσκολες και να μπορώ να τις εντάξω. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Πρόεδρε για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι έτσι απαντήσατε, έστω και αν είναι τεχνική η απάντηση και όχι πολιτική, νομίζω ότι δώσετε μια απάντηση ε, στην κυρία ε, Αμίτσι και νομίζω ότι έτσι μπορούν να ξεκαθαριστούν και οι πολιτικές αμφιβολίες. Ε, στο άρθρο 25 ε, γίνεται λόγος ε, για την αξιολόγηση και μάλιστα στο εδάφιο 3 του 25 αναφέρεται ότι υπό το φως των διαδικασιών αυτών η Κομισιόν μέχρι τις 30 Απριλίου του 2021 θα πρέπει να υποβάλει σύσταση συμμόρφωσης με το άρθρο 218 Περιμένω λοιπόν τις τροπολογίες σας. Ε, ευελπιστώ ότι θα μπορώ να τις εντάξω, να είναι εύκολες τροπολογίες και να μην μου δημιουργήσουν δυσκολίες. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ και να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη, την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη 5η Απριλίου, ε, μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες, τις οποίες παρακαλώ να υποβάλλετε στα αγγλικά. Προχωράμε τώρα στο επόμενο σημείο. Είναι παρουσίαση της Κομισιόν για την πρότασή της όσον αφορά την προστασία των ε, ατόμων ε, σε σχέση με τα ε, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών για την κατάξυση του κανονισμού 45-2001 και της απόφασης 1247-2002. Η πρόταση αυτή ε, αφορά ε, όλα τα θεσμικά ε, όργανα και οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες κτλ. και αφορά την συμμόρφωση με, την, με το κείμενο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εγκρίναμε την προηγούμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ως Πρόεδρος ότι είναι για μία ακόμα πρόταση της Κομισιόν που δεν συνοδεύεται από εξέταση επιπτώσεων και ε, να σας πω ε, ότι έχω την εντύπωση, για αυτή είναι προσωπική μου αίσθηση, ε, ότι φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και εγώ δεν θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό κάνουμε καλύτερη νομοθέτηση. Ωστόσο, θα δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στην Κομισιόν να παρουσιάσει την πρόταση και μετά στους εισηγητές, σκιώδης και οποιονδήποτε άλλον θέλει να πάρει τον λόγο έτσι ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων επί της προτάσεως. Ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Μίκο από την Κομισιόν. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σύντομα, η πρόταση αυτή της Κομισιόν παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της οικονομίας των δεδομένων τον Ιανουάριο και φυσικά προκύπτει από την έγκριση του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων και την αστυνομική οδηγία πέρσι. Λοιπόν, αυτό το νομοθέτημα μαζί με τον κανονισμό περί ηλεκτρονικής ε, ιδιωτικότητας ολοκληρώνει ένα τοπίο προστασίας δεδομένων ε, για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η ευθυγράμμιση αυτή με τον Γενικό Κανονισμό ε, ήταν απέτηση του κανονισμού και βεβαίως ε, απέτηση ήταν να εφαρμόσουμε τον νέο το νέο κανονισμό παράλληλα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολύ στενή πρόθεσμη, γιατί χρειάζεται να δοθούν και κάποιοι μήνες για να προετοιμαστούν τα θεσμικά όργανα μέχρι τον ε, Μάιο. Οι αρχές ε, εδώ πέρα που μας καθοδηγούσαν ήταν οι εξής. Ε, πρώτα απ' όλα όπως ε, σωστά αναφέρατε, πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τους κανόνες ε, στο μέγιστο δυνατό με τον γενικό κανονισμό. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για τον εθνικό δημόσιο τομέα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα. Νομίζω αυτό είναι το βασικό αυτής της ε, πρότασης. Και θα έχουμε άρα προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό ή αλλιώς έχουμε διοικητικά πρόστιμα. Πρέπει λοιπόν επίσης να δούμε το τι σημαίνει η συνθήκη της Λισαβόνας και όσον αφορά το μοντέλο της διακυβέρνησης πρέπει να αναγνωρίσουμε στο νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο την σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μετά με βάση τον τρέχοντα κανονισμό είναι πως είτε θα ευθυγραμμίσουμε τους υφιστάμενους κανόνες με τον κανονισμό τροποποιώντας δηλαδή τους υφιστάμενους κανόνες για να πούν κάποιες νέες έννοιες ε, προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό ήδη ή τα διοικητικά πρόστιμα. Έχουμε παρόλα αυτά διατηρήσει κάποιες ε, υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού 45-2001 όταν έχει αποδειχθεί ότι έχουν κάποια αξία. Και βεβαίως ε, αυτό το αφήνουμε και στην κρίση των αρμοδίων προστασίας ε, προσωπικών και υπάρχει και κάποια ευελιξία στα κράτη-μέλη και εκεί πέρα καθορίζουμε τους κανόνες για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε τα πράγματα με τον ε, Γενικό Κανονισμό, λαμβάνοντα υπόψη σε κάποιε περιπτώσει τι ιδιαιτερότητε, αποφεύγοντα την κριτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, και έχοντας ε, βεβαίως και κάποιες ε, πρωτοπόρες έννοιες όπως τα διοικητικά πρόστιμα και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Επόπτη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Και πάλι λοιπόν ε, θα προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν για να αφήσουμε λίγο χρόνο για να εφαρμόσουμε τον κανονισμό στο Συμβούλιο. Σκοπεύουμε λοιπόν να έχουμε τρεις αναγνώσεις ε, και μέχρι το τέλος του έτους ε, να εγκριθεί το νομοθέτημα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω χωρίς να πω πολλά πριν δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια να μην ευθυγραμμίζουμε μόνο τους κανόνες ε, αλλά με το να το κάνουμε αυτό να δίνουμε στα κράτη-μέλη το καλύτερο παράδειγμα για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πακέτο αυτό. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Ένστα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, ο κανονισμός είναι η εφαρμογή του πακέτου και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις λοιπές υπηρεσίες αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και βέβαια στο EDPS ε, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και τον οποίο ε, στηρίζουμε. Να πω πρώτα απ' όλα ευχαριστώ μετά την πρώτη συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε στενά. Έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε με την εφαρμογή ενός πακέτου και θα πρέπει ακριβώς να δούμε και με την οδηγία και με τον βασικό κανονισμό πώς θα παραμείνουμε σε μία γραμμή, να μην έχουμε επικαλύψεις. και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Αυτό στο οποίο ασκούμε κριτική είναι για νιωστή φορά ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου. Θέλουμε μια τέτοια αξιολόγηση και ζητάμε από την Κομισιόν να την κάνει για να πάμε έτσι στις διαβουλεύσεις. Ήδη Είπαμε πολλά πράγματα στις διαπραγματεύσεις, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Και εγώ αυτή την άποψη έχω έτσι ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή από το Μάιο του 2018. Νομίζω γι' αυτό πρέπει να κάνουμε γρήγορα τις συναντήσεις των σκιωδών πριν καταλήξουμε στην έκθεση και τις τροπολογίες. Πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Το πρώτο, να δούμε πώς ε, συνδέεται το θέμα αυτό με άλλες οδηγίες και κανονισμούς ή ε, privacy παραδείγματος χάρη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεύτερον, πρέπει να μιλήσουμε για το πεδίο εφαρμογή. Είναι μια γκρίζα ζώνη όταν μιλάμε για τα αποκεντρωμένα όργανα. είδαμε πως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν ε, κάποιες υπηρεσίες που έχουν δικό τους καθεστώς ε, προστασίας ε, δεδομένων. Τι κάνουμε εκεί με αυτή την τράπεζα δεδομένων όπως και με άλλες άλλωστε. Ζητήσαμε μία εικόνα από την ε, Κομισιόν για το πώς έχουν τα πράγματα με τους κανονισμούς ε, προστασίας δεδομένων. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, μεγάλα κενά εδώ πέρα, τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα δικαιώματα των υποκειμένων εδώ πέρα. Είναι σαφές, αλλά υπάρχουν και οι περιορισμοί που είναι οι λεγόμενοι εσωτερικοί κανονισμοί που δεν μας ικανοποιούν ιδιαίτερα, θεωρούμε ότι καλύτερο είναι να ρυθμίζονται τα πράγματα νομοθετικά. Εντάξει, αν είναι καμία μονομένη περίπτωση να το συζητήσουμε. Το EDPS για μας πάρα πολύ σημαντικός, ε, ο επόπτης ε, προστασίας δεδομένων πρέπει να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα και αρμοδιότητες σε σχέση με το Συμβούλιο και τον Επόπτη Θέλουμε έναν ισχυρό επόπτη ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του σωστά. Διαδικασία θέσης ε, σε εφαρμογή. Θα θυμόμαστε ήδη από τον επόπτη. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Ε, τέλος πάντων δεν είναι όλα αυτά τα οποία είχα να πω, αλλά είναι η πρώτη συζήτηση και χαίρομαι για την συνεργασία με τις ομάδες και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Άλμπρεχτ που είναι σκιώδης ηγετής για τους πράσινους. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που αρχίσαμε να ομαλά να εξετάζουμε αυτή την επιτροπή, την ε, πρόταση που επί της ουσίας ε, οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι που ήδη έθιξε η συγγετρία και που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερο προβληματικό, όπως είπε και η συγγετρία, ως προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γιατί στο Γενικό Κανονισμό αποφασίσαμε ως νομοθέτες ο κανονισμός 2001-145 να αφορά όλα τα δεδομένα που επεξεργάζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα. Οι οργανισμοί καλύπτονται δηλαδή. Κάτι που δεν ίσχυε στο κανονισμό 145 ε, του 2001, αλλά εμπίπτει στο Γενικό Κανονισμό της Προστασίας Δεδομένων. Είπαμε στο Γενικό Κανονισμό ότι ο κανονισμός αυτός θα εφαρμόζεται σε φορείς, οργανισμούς και θεσμικά όργανα. Και υπάρχει και ένας πολιτικός λόγος, μια πολιτική αιτιολόγηση για τη διεύρυνση αυτή του πεδίου εφαρμογή. Και ο λόγος είναι ότι καταρχήν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ζητήσαμε να έκαθεν οριζόντιες προδιαγραφές για την προστασία δεδομένων, εξού και ο γενικός κανονισμός της προστασίας των δεδομένων. Και δεν μας ε, άρεσε και πολύ που έπρεπε να συμφωνήσουμε για ένα ειδικό μηχανισμό για τις τηλεπικοινωνίες ή τα δεδομένα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Γιατί εμείς θέλαμε από την αρχή να το συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε μας άρεσε που έπρεπε να συμφωνήσουμε για μια ειδική οδηγία για την αστυνομία, την επιβολή νόμου και το δικαστικό κλάδο. Εν πάση περιπτώσει, σεβαστήκαμε αυτή την ε, ε, επιθυμία, αλλά αποφασίσαμε ότι ο Γενικός Κανονισμός θα είναι το ενιαίο όργανο που θα καλύπτει όλα τα θεσμικά όργανα, τους κοινοτικούς φορείς και τους ε, ενωσιακούς οργανισμούς. Συμπεριλάβαμε δηλαδή και τους οργανισμούς. Και το κάναμε αυτό γιατί αυτή τη στιγμή στον τομέα επιβολής ε, νόμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες διαφορετικά πρότυπα και προδιαγραφές. Κάθε σύστημα πληροφοριών, κάθε ε, φορέας, κάθε θεσμικό όργανο, κάθε οργανισμός εφαρμόζει τα δικά του πρότυπα και τις προδιαγραφές. Ιδιαίτερα ε, οι οργανισμοί ως προς τα συστήματα που έχουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν ε, σε ένα ενιαίο πακέτο, σε μια ενιαία δέσμη προδιαγραφών για να έχουμε ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών που θα εξυπηρετεί και την ασφάλειά μας και καλύτερη συνεργασία στον κλάδο και ταυτόχρονα ενώ απαιτούμε από τα κράτη μέλη κάτι τέτοιο, οποιαδήποτε σύστημα πληροφοριών ή οποιαδήποτε οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικό και κεκτημένο οι προδιαγραφέ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν νομίζω ότι στέκει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα τα κράτη-μέλη ήταν υπέρ τη συμπερίληψη όλων των θεσμικών αυτών φορέων και των ε, ενωσιακών οργανισμών στο Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων. Τελικά εμείς ε, στο Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε να δώσουμε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επεξεργαστεί την ε, ειδική βάση δεδομένων για τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασία Δεδομένων και, και το νέο συσταθέν Συμβούλιο Προστασία δεδομένων. Αλλά θέλουμε κάποιε οριζόντιε προδιαγραφέ και πρότυπα που θα ισχύουν για όλου του ε, κοινοτικού φορείς και του ε, οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σαφέ αίτημα και θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε του οργανισμού και τα συστήματα πληροφοριών ε, στο, στο πεδίο εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού, ώστε να έχουμε πραγματικέ ενιαίε, κοινέ προδιαγραφές, όπως χρειάστηκε να κάνουν τα κράτη-μέλη ε, ως προς την σχετική οδηγία και τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Άλμπρεχτ. Δεν ε, ζήτησε κάνει άλλο συνάδελφο το λόγο, οπότε θα το ξαναδώσω ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει, γιατί τέθηκαν ερωτήσεις για τον ορισμό των άλλων γραφείων και το σαφές αίτημα για εναρμόνιση των προδιαγραφών σε όλους ε, τους κοινοτικού θεσμούς, φορείς και οργανισμούς. Επίσης, τι θα γίνει με την ε, δυνατότητα επιβολής προστήμων. Πώς θα το οργανώσουμε αυτό. Και επαναλαμβάνω το, ε, το αίτημα της κυρίας Έρνστ να εκπονηθεί μελέτη επιπτώσεων. Παρόλο που ξέρουμε ότι θέλουμε ταχεία διαδικασία ώστε όλα να εφαρμοστούν ήδη από τις αρχές του 2018. Κύριε Μικόλ, θα μπορούσατε να κάνετε κάποια σχόλια ή να δώσετε απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη μελέτη αντικτύπου. Ελήφθη απόφαση να μην καταρτιστεί η μελέτη αντικτύπου λόγω του περιορισμένου πεδίου εφαρμογή τη σχετική πρόταση και επειδή πρόκειται για ευθυγράμμιση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Εκπονήθηκε μία μελέτη που ολοκληρώθηκε και είναι και διαθέσιμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις διάφορες βάσεις δεδομένων. Οι περισσότερες ε, βάσεις δεδομένων εμπίπτουν σε έλεγχο που δεν είναι κοινοτικός είναι οι εθνικές αρχές αυτές που είτε υποβάλλουν ε, δυνάμει του Γενικού Κανονισμού ε, είτε της ε, οδηγίας για την αστυνομία, τα σχετικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, εδώ μιλούμε για δύο-τρεις οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής σχετικής πρότασης. γιατί γνωρίζουμε ότι πολύ πρόσφατα έχουν υιοθετηθεί τα σχετικά συστήματα, οπότε και μια και πρόκειται για νεοσυσταθέντες οργανισμούς, κρίναμε σκόπιμο να μην ε, ε, ξαναρχίσουμε συζήτηση από τώρα. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, αποτέλεσαν το αντικείμενο εκτενού συζήτηση και στην, εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρόκειται για μια τελείω πρωτοπόρα καινοτόμα προσέγγιση. Να δίνουμε δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Επόπτη αρμοδιότητα επιβολή προστήμων στου κοινοτικού φορεί ε, και θεσμικά όργανα. Βέβαια, έχουμε περιλάβει και μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων ώστε πραγματικά να είναι ίστατη λύση αυτά τα πρόστιμα και να μην επηρεάζουν δυσανάλογα τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Φορέων και ιδιαίτερα των μικρών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα κονδύλια που θα εισπραχθούν από τα πρόστιμα αυτά, όπως αναφέρεται και στο κείμενο, ε, θα τροφοδοτήσουν το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, περισσότερο αυτή η πρόταση έχει συμβολική αξία ε, και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που δίνουμε στην προστασία των δεδομένων στους κοινοτικού φορείς και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα και πάλι το λόγο στην κυρία Έρνστ, την εισηγήτριά μας, που ενδεχομένω ε, θα έχει κάποιε επιπλέον απορίε μετά τα σχόλια τη επιτροπή δεν συμφωνούμε με αυτά τα οποία μόλις ε, είπατε. Εμείς παραμένουμε στην απέτησή μας. Εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά με βάση μια παρουσίαση για υπηρεσίες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες, για να έχουμε εικόνα γιατί ακριβώς μιλάμε τελικά, έτσι, αυτό. Αυτά λοιπόν. Είμαι πολύ αισιοδόξη πάντως. Ευχαριστούμε κύριε Άρνστ. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, νομίζω ότι μη τι άλλο, θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο σχετικά νέοι κανόνες για τους οργανισμούς ευθυγραμμίζονται όντως με την ισχύουσα δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων. Οπότε ίσως καλό θα ήταν να γίνουν όλα αυτά εκ παραλίλου με την ανάλυση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν είναι μόνο τεχνικά αυτά τα θέματα, δεν είναι απλώς θέματα ευθυγράμμισης. Θα χρειαστούν και πολιτικές συζητήσεις για να δώσουμε πραγματικά το καλό παράδειγμα και για τα κράτη-μέλη. Μια χαρά που τα πάμε με το χρόνο σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έχουν έρθει οι αρμόδιοι. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Σδεχόφσκι για το σχέδιο συμφωνίας ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας με θέμα τους συμπληρωματικούς κανόνες ε, για τα μέσα χρηματοδοτικής στήριξης για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις ως τμήμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020. Μια και ο κύριος Δεχόφσκι κολλείεται σήμερα θα μας παρουσιάσει τη θέση του, το σχέδιο έκθεσης, ο κύριος Κοέλιος, τον οποίο και δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Στεχόφσκη, γιατί βρίσκεται στη Μάλτα σε συνεδρίαση του ΕΛΚ. Πάντως ο εισηγητής θέλει να υπογραμμίσει ότι το μέσο χρηματοδοτική στήριξη στο τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλεια, Σύνορα και Θεωρήσει για την περίοδο 2014-2020 είναι σημαντικό εργαλείο για να εξασφαλιστεί, υψηλό επίπεδο ασφάλεια στην Ένωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλού επίπεδου έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και αποτελεσματική επεξεργασία των θεωρήσεων στο χώρο Σέγγεν. Θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των συμμετοχών των χωρών του χώρου Σέγγεν και των συνδεδεμένων χωρών όπως είναι η Νορβηγία. Γιατί όχι μόνο θα πρέπει όλα τα κράτη να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συμβάλλουν και χρηματοδοτικά. Η πρόταση λοιπόν αυτή αφορά την Νορβηγία, που είναι συνδεδεμένη χώρα που συμμετέχει στο κεκτημένο του Σέγγεν και προσδιορίζει τον, τη συνεισφορά της Νορβηγίας στον, εσωτερικό, στον, στον προϋπολογισμό που είναι 19,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ε, για την ε, τροφοδότηση του Ταμείου Συντερική ασφάλεια. Ο εισηγητή ε, θεωρεί ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να στηρίξει την πρόταση, γιατί μέσω αυτού του χρηματοδοτικού μέσου θα έχουμε πιο αποτελεσματικό και ομοιόμορφο επίπεδο ελέγχου των εξωτερικών μα συνόρων και θα έχουμε καλύτερη επισκόπηση και επιτήρηση των συνόρων για να βλέπουμε ποιοι εισέρχονται και εξέρχονται από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο το θέμα της, του αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, για να είμαστε βέβαιοι ποιος εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια συζήτηση ε, να εξελίξει και θα πρέπει ε, να θέτουμε το ζήτημα όχι μόνο με τα κράτη-μέλη, αλλά και με συνδεδεμένες χώρες, με χώρες με τις οποίες έχουμε στενή συνεργασία. Και από αυτήν την άποψη είναι πολύ σκόπιμη και επίκαιρη έκθεση, γιατί δεν αφορά, επαναλαμβάνω, μόνο το θέμα του ελέγχου των εξωτερικών σύνορων, αλλά και το θέμα της ε, χρηματοδοτικής ε, στήριξης και χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Και από αυτήν την άποψη είναι πολύ σημαντικό το θέμα και η έκθεση. Ε, πολύ συχνά έχουμε εκθέσεις που απαιτούν ε, ταχεία διαδικασία. Ισχύει και για αυτή την έκθεση και εδώ η προθεσμία για τις τροπολογίες έχει οριστεί για την επόμενη Τετάρτη, 5 Απριλίου του 2017, στις 12 το μεσημέρι, τότε λίγη προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών στα αγγλικά και σε αντίθεση με άλλες εκθέσεις μου λέει τώρα η γραμματεία ότι δεν χρειάζεται να υποβάλλετε μόνο στα αγγλικά τις τροπολογίες σας μπορείτε να τις υποβάλλετε σε ό,τι γλώσσα θέλετε και μια και έχουμε κερδίσει αρκετό χρόνο, να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα γίνει τέλη Απριλίου, 24 ή 25 Απριλίου του 2017 και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για το Μάιο 2017. Δεν βλέπω όμως κανέναν αρμόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίμαχο το θέμα. Οπότε μπορούμε κάλλιστα να περάσουμε στο επόμενο. Πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση ενταλμάτων δέσμευσης και δίμευσης το προτινόμενο αυτό μέσο θα αντικαταστήσει την ε, ισχύουσα Συμφωνία Πλαίσιο του Συμβουλίου 2006-783 για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε εντάλματα δίμευσης και την απόφαση πλαίσιο 2003-577 για τα εντάλματα δέσμευσης. Να σας υπενθυμίσω ότι το 2014, η Οδηγία 2014-42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε με θέμα τη δέσμευση και δίμευση ε, περιουσιακών στοιχείων ε, που είναι αντικείμενα προϊόντα εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οδηγία Ενορμόνησης ε, προέβλεψε κάποιους κοινούς κανόνες και προδιαγραφές για δημεύσεις στο ποινικό δίκαιο, καθώς και κάποιες μορφές παρατεταμένων δημεύσεων, εκτεταμένων δημεύσεων και δημεύσεων ε, χωρίς να έχει προηγηθεί κατά δίκη σε δύο περιπτώσεις εξαφάνισης και ασθένειας. Ε, προτινόμενος κανονισμός από την άλλη πλευρά προβλέπει αμοιβαία αναγνώριση τέτοιων μέτρων του ποινικού δικαίου που είναι επίση εκτό ε, του πεδίου της εναρμόνισης. Να σα υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση στο ποινικό δίκαιο, έχουμε ένα άλλο πρόσφατο νομοθετικό μέσο, την Οδηγία 2014-41 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης. Και η οδηγία τότε είχε κλειφθεί ως πρότυπο πλαίσιο για την μελλοντική αμοιβή αναγνώριση σε θέματα ποινικού δικαίου, γιατί υπήρχε συνένεση μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων τότε, ακόμη και για την συμπερίληψη ε, μίας, ε, ενός λόγου μη αναγνώρισης των πολιτικών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ακριβώς επειδή έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο, δεν έχει προφτάσει να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά η συγγήτριά μας είναι εδώ. Μια και είναι παρούσα όμως η συγγητριά μας, η κυρία Γκρισμπέκ, μπορεί να κάνει αυτή την αρχή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πάντως ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η Κομισιόν. Δηλαδή πρώτα να παρουσιάσει η Κομισιόν ε, τις ε, γενικές ε, γραμμές, αλλά μια και είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, νομίζω ότι καλό είναι να μην αντιστρέψουμε την σειρά. Εγώ μπορώ, αν θέλετε, να μιλήσω, μπορώ να πάρω το λόγο τώρα, αλλά νομίζω ότι από παιδαγωγική, ας πούμε, απόψεως, θα ήταν καλύτερα να μιλήσει πρώτα η Κομισιόν. Και μάλιστα λείπουν και οι σκιώδεις Κανένα σκιώδη δεν είναι. Ίσως τότε, λέει η Πρόεδρο, είναι καλύτερα να διακόψουμε για λίγο, έτσι ώστε πράγματι και η Κομισιόν και οι σκιώδη να είναι εδώ. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. 9 λεπτών, είναι 9 και 51, στις 10 να είμαστε ξανά εδώ. So you can have a coffee, yes. Οπότε, συναδελφοί, αφού έχω κάνει ήδη την εισαγωγή για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την αμοιβαία αναγνώριση για τις αποφάσεις ε, δήμευσης και κατάσχεσης ε, κάθισαμε άλλα τρία λεπτά μια που έχουμε κάνει λοιπόν την εισαγωγή θα δώσω απευθεία τον λόγο στην Κομισιόν και μετά στους εισηγητές. Ε, κύριε Σρέντερ, έχει τον λόγο. Κυρία Σρέντερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ μου δίνετε τον λόγο να παρουσιάσω την ε, πρότασή μας για την αμοιβή αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης Λοιπόν, έχουμε μια γενική εικόνα να σας δώσω. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο η δέσμευση στοιχείων ε, του εγκλήματος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο καταπολέμησης του εγκλήματος καθώς έτσι αφαιρούμε από τους εγκληματίες τα κέρδη του εγκλήματος και ταυτόχρονα παρέχει επιπλέον κονδύλια που επενδύονται στην επιβολή του νόμου ή σε άλλους σκοπούς ή και για κοινωνικούς σκοπούς. Η δέσμευση και δίμευση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό μέσο καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς διαταράσει τα έσοδα των ε, τρομοκρατικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια του 2015 τόνισε την ανάγκη του να αντιμετωπιστεί η χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας με τρόπο αποτελεσματικό και συνολικό, καθώς επίσης και την ανάγκη βελτίωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, δέσμευσης και δίμευσης. Επιπλέον, η Κομισιόν δεσμεύτηκε το 2016 ε, να καταπολεμήσει την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και επίσης αντιδρώντας ε, σε εκκλήσεις ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου όταν η οδηγία 1442 είχε εγκριθεί για να προετοιμάσουμε μια νέα νομοθετική πρόταση για την ομιλία αναγνώριση δέσμευσης και δημευσής. Αυτό κάναμε λοιπόν. Έχουμε τώρα αυτή την πρόταση που προτείναμε στα τέλη του 2016. Τα κύρια προβλήματα που διαπιστώσαμε προετοιμάζοντας αυτή την πρόταση είναι τα εξής. Πρώτον, υπήρχε υπάρχει ακόμα ανεπαρκής ανάκτηση των προϊόντων εγκλήματος σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Πάρα πολύ λίγα από αυτά δεσμεύονται και δημεύονται σε διασυνοριακές περιπτώσεις και σε αυτά σε μια κατάσταση στην οποία τα προϊόντα εγκλήματος ε, μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη. Για τους λόγους τώρα της ε, ανεπαρκούς ανάκτησης ε, βλέπουμε πως ε, υπάρχουν δύο αποφάσεις πλαίσιο το 2003 και 2006 στο πλαίσιο το νομοθετικό οι οποίες δεν καλύπτουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην νομοθεσία κάποιων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ορίζει κάποιους ελάχιστους κανόνες. Συγκεκριμένα η οδηγία του 2014-42 για τα προϊόντα εγκλήματος που αυτή ευκαιρία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία μέχρι το φθινόπωρο που μας πέρασε. Οπότε το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων αυτών είναι περιορισμένο και δεν καλύπτει πολλές ε, περιπτώσεις δίμευσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη που περιλαμβάνουν και την δίμευση μετά από καταδίκη. Αυτό ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι τα πισταποιητικά και οι διαδικασίες που αναφέρονται στα υψηλά μέτρα είναι πολύ περίπλοκα και αναποτελεσματικά. Και δεν υπάρχουν παραδείγματο χάρη προθεσμίες. Και τέλος υπάρχουν μέσα τρίτου πυλώνα που δεν είναι άμεσα εφαρμόσουμε και αφήνουν μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Οπότε, αυτό ήταν το πρώτο γενικό πρόβλημα. Το δεύτερο που βρήκαμε ήταν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπει αποζημίωση των ε, θυμάτων μέσω δίμευσης σε διασυνοριακές υποθέσεις. Οπότε έχουμε κάποια κράτη-μέλη όπου το κράτος μπορεί να δημεύσει για λογαριασμό των θυμάτων του εγκλήματος, αλλά όχι σε όλα τα κράτη-μέλη και η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει σε διασυνοριακές ε, υποθέσεις. Οπότε ε, θεωρούσαμε ότι έπρεπε και αυτό να καλυφθεί. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά στοιχεία. Πρώτον, πρόκειται για ένα μέσο αμοιβαίας αναγνώρισης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η απόφαση μιας δικαστικής αρχής ε, ενό κράτου μέλου θα αναγνωρίζεται και θα εφαρμόζεται από άλλο κράτο μέλο χωρί να αξιολογείται ξανά επί τη ουσία. Βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εναρμόνιση κανόνων. Είναι απλά ένας μηχανισμός διασυνοριακής συνεργασίας και καλύπτει όλα ακριβώ ε, τα μέσα που υπάρχουν. Τι είναι εκτεταμένη δίμευση, δίμευση ε, από τρίτους ε, και βεβαίως η πρόταση αυτή θα βελτιώσει το πλαίσιο με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα είναι μια πρόταση για κανονισμό. Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν προτείνει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο μέσο το προηγούμενο μέσα ήταν ε, αποφάσεις ε, πλαίσιο και το προηγούμενο που είχαμε ήταν η οδηγία για, την, για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα έρευνα. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε κανονισμό που θα ισχύει απευθεία, ε, θα παρέχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και δεν θα υπάρχουν προβλήματα μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ενώ η οδηγία ε, δίνει στα κράτη-μέλη κάποιο περιθώριο για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και άρα μπορεί να διαφέρει η νομοθεσία από τη μια χώρα στην άλλη και στην περίπτωση του κανονισμού δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο και επειδή μιλάμε για διασυνοριακές ε, διαδικασίες ε, δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει τέτοια διακριτική ευχέρεια. Οπότε είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή είναι η καλύτερη μορφή αυτού του μέσου σε αυτή την περίπτωση και θα υπάρχει έτσι σαφήνεια και δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή. Κατόπιν για το πεδίο εφαρμογής θα πηγαίνει πέρα από τις διαδικασίες πλαίσιο θα καλύπτει όλες τις μορφές ε, δίμευσης ε, που εναρμονίζονται στην οδηγία του 2014-42 δηλαδή παραδοσιακή δίμευση δίμευση από τρίτους ε, και εκτεταμένη επίσης ε, δίμευση και επίσης δίμευση χωρίς ε, καταδίκη δέσμευση χωρίς καταδίκη και θα καλύπτει βεβαίως και τις άλλες μορφές αρκεί να είναι εντός του πλαισίου ποινικών διαδικασιών. Οπότε εδώ εξετάζουμε τις ε, περιπτώσεις ε, ασυλίας όπου ο δράστης είναι άγνωστος ή όταν το δικαστήριο μπορεί να δεσμεύσει κάποια πράγματα όταν θεωρεί ότι είναι προϊόντα εγκλήματος ακόμα και αν δεν υπάρχει καταδίκη. Και επειδή μιλάμε βεβαίως για ποινική διαδικασία ισχύουν ε, και όλες οι δικλείδες ασφαλείας ε, που ισχύουν συνήθως. Ένα άλλο πλέον έκτημα είναι ότι προτείνουμε να εισαχθούν προθεσμίες για διαδικασίες δέσμευσης ε, που είναι κάτι το πιο κατεπήγον είναι πιο σύντομες οι προθεσμίες ενώ για αναγνώριση και εκτέλεση εντολής δίμευσης είναι πιο εκτεταμένες ε, και βεβαίως μετά εισάγεται και ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό, ένα έγγραφο το οποίο θα επιτρέψει γρήγορη και αποτελεσματική δράση και θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε η εκτέλους αρχή να μπορέσει να εκτελέσει την απόφαση. Τέλος, Υπάρχουν πολλές ε, διατάξεις στην πρόταση για την επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών που είναι ένας βασικός παράγων επιτυχίας ε, της αμοιβαίας αναγνώρισης και για τα δικαιώματα των θυμάτων που ανέφερα υπάρχει τώρα μια διάταξη που επιτρέπει στις ε, περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί μία εντολή αποζημίωσης ή ανάκτησης και σε ένα κράτος μέλος και έχουν δεσμευτεί κάποια πράγματα σε άλλο κράτος μέλος να υπάρχει ε, η δυνατότητα να έχει προτεραιότητα το ε, θύμα εναντί των υπολείπων για να λάβει ένα μέρος του ποσού το οποίο θα ανακτηθεί. Και τέλος να κλείσω για το εάν ε, προστατεύονται παρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο κανονισμός λοιπόν που προτείνεται θα καλύπτει μόνο τις εντολές που εκδίδονται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, οπότε ισχύει οτιδήποτε ισχύει για τις ε, ποινικέ διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη που αναφέρεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο ποινικό της ε, τμήμα, άρθρο 6 παραγραφός 3 δηλαδή, επιπλέον την ε, σχετική κοινοτική νομοθεσία που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και τις έξι οδηγίες που έχουμε τώρα για τα δικονομικά δικαιώματα, δηλαδή δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση, πρόσβαση σε ε, δικηγόρο, το τεκμήριο της αθωότητας ε, και οικονομικές εγγυήσεις για παιδιά και νομική αρρωγή. Λοιπόν, δεν ε, θεωρήθηκε επίσης αναγκαίο να περιλάβουμε συγκεκριμένη αιτιολόγηση απόρριψης με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς μιλάμε για ποινικό δίκαιο ε, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να, θα μπορούσε να υπάρχει ευρύτατη ερμηνεία από τους δικαστές και να υπάρχει άρα πρόβλημα με την αμοιβαία αναγνώριση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, για όλες αυτές τις πράγματι λεπτομερείς ε, ε, παρουσιάσεις που μας κάνατε. Θα ήθελα τώρα να, λόγω τον, να δώσω τον λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ανταλή Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σρέντερε για την ε, παρουσίαση που έκανε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν ε, μία παρουσίαση λεπτομερής αλλά όχι υπερβολικά τεχνική για ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό σε ποινικό επίπεδο βεβαίως αλλά και γενικότερα ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και αγγίζει πάρα πολύ ε, τους ε, ε, πολίτες της Ευρώπης αλλά και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές των κρατών στην προσπάθειά τους ας πούμε να συγκρατήσουν την τρομοκρατία και να την αποτρέψουν στην, στο ξεκίνημα τους. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν τον προηγούμενο Δεκέμβρη που μας δίνουν την ε, δυνατότητα ε, να αποκτήσουμε ε, τρόπους καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αλλά βεβαίως και του οργανωμένου εγκλήματος. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε άμεσα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει από το ξεκίνημα του να καταπολεμηθεί ε, με ε, τρόπο αποτελεσματικό. Ήδη από το 2015 και εντονότερο το 2016 αυτή η δαμόκλειος πάθη της ε, τρομοκρατίας είναι πλέον τόσο σημαντική που πρέπει να μας οδηγήσει σε καλή συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το είπατε κι εσείς άλλωστε έμεσα, για να κατα για να μπορέσουμε να προλάβουμε ε, τα τρομοκρατικά σχέδια μέσω της ε, μείωσης ε, της χρηματοδότησης πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να μειώσουμε τις πηγές χρηματοδότησης και επομένως την χρηματοδοτική ικανότητα ε, ε, που έχουν οι ομάδες αυτές. Δεν το είπε ξεκάθαρα η Κομισιόν, αλλά πάντως ανέφερε ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν να αποζημιωθούν αποτελεσματικά και σωστά τα θύματα όταν επιτρέπεται αυτό από την Εθνική Νομοθεσία, αλλά διεφάνει επίσης ότι θα χρήματα αυτά αυτά θα αποτελέσουν επιπλέον κονδύλια τα οποία μπορούν ε, να επανατοποθετηθούν ε, σε όλες τις δραστηριότητες ε, πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Επομένως το κείμενο και το σχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης δέσμευσης και δίμευσης όλων αυτών των χρηματοδοτικών πηγών έτσι ώστε να αποκοπεί η χρηματοδοτική ικανότητα τροφοδότησης α πούμε με αυτών των ε, τρομοκρατικών ε, ομάδων. Ε, θα ήθελα να μπορώ να είμαι απολύτως βέβαιη όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, παρόλο που είναι δύσκολα. Είχα κάποια ερωτήματα, αλλά με απαντήθηκαν ήδη από την αρχική σας παρέμβαση, κυρίως όσον αφορά ε, την ε, αιτιολόγηση απόρριψης ε, βάσει επιχειρηματολογίας σχετικής με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Απαντήσατε ήδη στο θέμα αυτό. Μία πρώτη παρατήρηση μπορώ να κάνω. Εκτιμώ ιδιαιτέρως το μέσο το οποίο επελέγει η Κομισιόν προτείνει κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση αυτών των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό ε, νομικό ε, εργαλείο και δείχνει ότι ε, υπάρχει βούληση για γρήγορες διαδικασίες ε, και επομένως ε, μιλάμε για ποινικέ διαδικασίες και ε, άρα είναι ένα μέσο ο κανονισμός που μας δίνει περισσότερες δυνατότητες. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να είμαστε απολύτως σαφείς και συγκεκριμένοι όσον αφορά το μέσο το οποίο θα αποφασιστεί τελικά από, τις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα πρέπει να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Μας υποχρεώνει δηλαδή όλους να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Επίσης, ε, μια διευκρινιστική ερώτηση, όχι πολύ μεγάλη εμβέλεια. μήπως η Κομισιόν θα μπορούσε ε, πιο ξεκάθαρα να αναφέρει ε, τις διευκρινήσεις ή τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στις δύο υφιστάμενες οδηγίες ε, Ποιε είναι οι τροποποιήσεις δηλαδή που γίνονται με αυτόν τον νέο κανονισμό. Αλλά βέβαια θα το δουλέψουμε το τεχνικό αυτό κείμενο με τους ε, σκιώδει συγητέ. Μπορεί να είναι τεχνικό αλλά είναι και ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ Ναταλή. Ναι βεβαίως ε, είναι τεχνικό κείμενο αλλά συμφωνώ μαζί σου όταν λες ότι όλοι οι πολίτε της Ευρώπη θέλουν να κοπεί η χρηματοδοτική τροφοδότηση των ε, ε, ομάδων, των τρομοκρατικών ομάδων και επομένως η δέσμευση και η δίμευση ε, αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε ότι διασφαλίζονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ο σεβασμός τους πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους σκιώδους, σκιώδεις εισηγητές εφόσον είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε κύριε Γκρίσμπεκ και εγώ, κύριε και εγώ προσβλέπω σε, σε συνεργασία στενή μαζί σας αυτό το σημαντικό θέμα και μια και η διαδικασία έγκρισης ενός κανονισμού επίσημα βρίσκει σύμφωνο γιατί άλλες είναι οι συνέπειες του κανονισμού και μας εξήγησε το σκεπτικό της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρετίζουμε την πρόταση. Και είναι θετική η πρόταση, αν σκεφτούμε ότι 8,1% των ε, περιοσιακών στοιχείων ε, που είναι προϊόντα εγκλήματος εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για να προκαλούν περισσότερες ζημίες ακόμη στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν φυσικά να εξασφαλίσουμε και να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό όμως το τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης τα δημευθέντα σε άλλο Ευρωπαϊκό κράτο περιουσιακά στοιχεία, μετά την διαδικασία αμοιβαία αναγνώρισης θα πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα αποζημίωση ή επιστροφής στα θύματα και θα έχουν προτεραιότητα τα συμφέροντα του κράτου μέλους έκδοσης και εκτέλεσης. Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να οικοδομήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη Ε, γιατί και αυτά θα υποφεληθούν από τις αποζημιώσεις. Μία τέτοια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ακόμη και αν ε, έχει ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος με διαφορετικές συνέπειες, αλλά θα πρέπει ε, να τηρούμε την αρχή του ουδής δικάζειν, εμπί Σε ό,τι αφορά τις, τα εντάλματα δέσμευσης και δίμευσης, θα πρέπει να έχουμε σαφείς προθεσμίες ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές διασυνοριακές διαδικασίες, γιατί τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται γρήγορα, γι' αυτό και θέλουμε βραχίες προθεσμίες που θα είναι, θα πιο θα είναι και πιο αποτελεσματικές. Ελπίζω να το λάβετε υπόψη. Προκειμένου να γίνει βέβαια αναγνώριση και εκτέλεση τέτοιων ενταλμάτων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν όπου δει, όπως είπατε και εσείς, τα στοιχεία αυτά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Και μια και πρόκειται για κανονισμό, ελπίζω μετά την αργότερη αυτή προσπάθεια που θα κάνουμε να συγκεντρώσουμε και μεγάλη πλειοψηφία ε, για να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα προς τους πολίτες ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για τα συμφέροντά τους. Σας ευχαριστούμε κύριε Πάβελ. Επόμενος ομιλητής είναι ομιλήτρια, η σκευδεσηγήτρια κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Σνέρντερ αλλά και την Ναταλή για τις εισηγήσεις που μας έκαναν. Εγώ προέρχομαι από την Ιταλία και κατανοώ ε, την μεγάλη χρησιμότητα ενός ε, μέσου ε, που θα έχει αυτό, αυτά τα δεσμευτικά χαρακτηριστικά του κανονισμού. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο καταπολέμησης της μαφίας στην χώρα μου. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ε, γιατί ε, εμείς είχαμε λάβει κάποια μέτρα πριν αρχίσει ε, η οι τρομοκρατικές επιθέσεις γιατί στην χώρα μου η καταπολέμηση των μαφιόζικων ας πούμε εταιριών καταπολεμούνται ε, ε, περνάει μέσα από την ε, δέσμευση και την δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τέτοιου είδους αποφάσεις μπορεί να έχουν πολύ αποτελεσματική επίπτωση στην τρομοκρατία γιατί η τρομοκρατία είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει ακόμα καλά καθοριστεί στα νομοθετικά μας συστήματα. Ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη βεβαίως ε, και τα δικαιώματα των μέσων, των μελών μάλλον των δρομοκρατικών ε, ομάδων. Ε, θα πρέπει να μελετήσουμε καλά το θέμα ε, όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση δεσμεύσεων και δημεύσεων που δεν βασίζονται σε ποινικέ αποφάσεις και που βασίζονται στην οδηγία 42 του 2014. Κατά αυτή την έννοια, όσα μας είπε η κυρία Σρέντερ σήμερα, είναι πολύ σημαντικά. Ξαναναφέρομαι όμως αυτά γιατί πολλές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ε, μαρτυρούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, κάποιοι κίνδυνοι εγγενείς στις αποφάσεις δέσμευσης και δίμευσης ε, με την έννοια ότι μπορεί τέτοιες αποφάσεις να παραβιάζουν κανόνες που προβλέπονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο ρόλος ε, των σκιωδών εισηγητών ε, είναι, ε, και αυτό θα κάνω και εγώ ως σκιώδης, να μελετήσει σε βάθος και να κατανοήσει τα προβλεπόμενα και εγώ αυτό θα πράξω. Θα προσπαθήσω να δω σε βάθος ε, τα προβλεπόμενα έτσι ώστε να μην υπάρχει αντίθεση ή αντίφαση ε, με, τις, ε, με την ομολογία καθώς επίσης και με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 42 του 2014, ε, εάν ε, υπάρχουν ισχυρές ε, ενδείξεις βάσει έρευνας και αν υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και εάν οι αρχές δεν έχουν σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τότε ε, θα έπρεπε και πρέπει να απορριφθεί ε, η απόφαση δέσμευσης ε, και δίμευσης. Αυτού του είδους τα στοιχεία θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος και αυτό θα κάνω και εγώ. Ευχαριστώ την Ναταλή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράου είναι ο επόμενος συμμιλητής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως έλεγε και η συνάδελφος Σπινέλη και εγώ γνωρίζω την Ιταλική εμπειρία. Ε, στην Ιταλία λοιπόν αυτό το εργαλείο ε, ήταν πραγματικά ε, ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτή η δυνατότητα δέσμευσης και δίμευσης προϊόντων ε, ε, εγκληματικών ενεργειών από την αρχή μέχρι το τέλος της ε, διαδικασίας ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα γιατί από την αρχή της διαδικασίας μέχρι το τέλος ενδεχομένως τα προϊόντα αυτά εξαφανίζονται και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Θεωρούμε ότι τέτοιες αποφάσεις είναι σωστές και θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό μάλιστα ήταν και πάγιο αίτημα των ε, οργανώσεων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και των μαφιών ε, στην ε, Ιταλία. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ε, ενδιαφέρει και μας πάρα πολύ και μάλιστα αποτέλεσε και αντικείμενο ε, ψηφίσματος ιδίας πρωτοβουλίας ε, στο Κοινοβούλιο. Το εργαλείο της οδηγίας, του κανονισμού, συγγνώμη, βεβαίως μας βρίσκει απολύτω σύμφωνος γιατί είναι συγκεκριμένο και δρά γρήγορα. Και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής μας βρίσκει θετικούς. Η δυνατότητα άμεσης δέσμευσης και δίμευσης πριν από την τελεσίδικη ποινική καταδίκη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, βεβαίως εδώ ε, μιλάμε ε, για την δυνατότητα των κρατών μελών να αντιταχθούν στην απόφαση εκτέλεσης. Βεβαίως το παρεμίπτον ερώτημα είναι αν τα κράτη-μέλη θα σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και εάν απαντήσουμε θετικά και στα δύο ερωτήματα, τότε πραγματικά το εργαλείο θα έχει ε, συγκεκριμένη εφαρμογή. Το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος και όχι μόνο της τρομοκρατίας ε, ε, είναι πλέον παγκοσμιοποιημένο και μάλιστα το οργανωμένο έγκλημα έχει παγκοσμιοποιηθεί με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του εμπορίου και ξέρουμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σε αυτήν την ταχύτατη εξάπλωση έστω και αν ε, ε, ο κατάλογος των αδικημάτων ε, είναι πάρα πολύ μεγάλος, τον είδαμε και πραγματικά είναι ε, ενδελεχής και προβλέπουν και μέγιστη ποινή ας πούμε τριών ετών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για την πρώτη της παρουσίαση και ευχαριστούμε πολύ για την εισηγήτρια την οποία προτιθέμεθα να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη εργασία που έχει αναλάβει. Ευχαριστώ. Thanks Σας ευχαριστούμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το έργο σας, γιατί ακριβώς οι διαφορετικοί κανόνες που έχουμε στα κράτη-μέλη είναι απόρρια των διαφορετικών μας εμπειριών και επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τις κοινωνίες μας. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να ζητήσουμε κάποιους κοινούς κανόνες που θα γίνονται σεβαστοί από όλου και θα είναι και αποτελεσματικοί ταυτόχρονα. Επίσης το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μόλις πριν από δύο εβδομάδες είχαμε δημόσια ακρόαση με αστυνομικούς από πολλές χώρες που μας επισήμαναν ότι όλο και περισσότερες αξιόπινες πράξεις έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ενίσχυση της συνεργασίας προκειμένου να είναι αποτελεσματική και να μας επιτρέψει να αναχαιτήσουμε έστω και κάποιες μορφές εργανομένου κλίματος και τρομοκρατίας. Και πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εισηγήτρια πως θέλουν να προσθέσουν κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστώ να απαντήσω στις απορίες της εισηγήτριας. Ρωτήσατε ποιο είναι το βασικό πλονέκτημα της ε, νέας πρότασης σε σχέση με την απόφαση πλαίσιο. Ως προς τη μορφή αυτή είναι το μείζον πλονέκτημα, είναι δεσμευτικός ο κανονισμός και επίσης θα έχουμε ένα ενέο, ε, μια νέα νομοθετική πράξη που με συνεκτικό τρόπο θα καλύπτει και τη δέσμευση και τη δίμευση. Ε, επίσης, ε, εκτεταμένο πεδίο εφαρμογή πιο διαβριμένο σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό μέσο. Τα κράτη-μέλη, πολλά κράτη-μέλη τουλάχιστον, έχουν ε, ε, αντιληφθεί πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι τα εντάλματα δέσμευσης και δίμευσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό και ενίσχυσαν ε, τα εθνικά του συστήματος και είχαμε και την οδηγία φυσικά του 2014 που επίσης επέφερε κάποιο βαθμό εναρμόνισης. Οι προηγούμενες αποφάσεις πλαίσιο κάλυπταν την περίοδο 2003-2006. Ήταν αρκετά ξεπερασμένε. Πρέπει να προσαρμοστούμε στι νέε εξελίξει. Εξού και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Ε, οι προθεσμίε αναφέρθηκαν. Ε, μέχρι τώρα δεν είχαμε. Τώρα έχουμε τι τρίμερε προθεσμίε για τη δέσμευση και 30 και κάτι μέρε για τα εντάλματα δίμευση. Έτσι, ιδιαίτερα για τη δέσμευση, που σε διασυνοριακές διαδικασίες η άμεση αντίδραση έχει σημαντική, σημαντικό αποτέλεσμα προκειμένου να δεσμεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία πριν να προλάβουν οι εγκληματίες ε, να τα εξαφανίσουν. Και προβλέψαμε και κάποιες διατυπώσεις, κοινοποίησης και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό σας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, προβλέπουμε και δυνατότητες προσφυγής για, τους, ε, όσους έχουν πληγεί από αυτά τα μέτρα, που όντως ε, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στου στους πολίτες. Οπότε η πρόταση διευκρινίζει ότι τα 11 μέσα οι δικαστικές προσφυγές μπορούν να υποβληθούν μόνο στο κράτος έκδοσης, αλλά σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπεται η άσκησή τους και στο κράτος εκτέλεσης. Επίσης προβλέπονται κοινοποιήσεις ε, για να γνωρίζει ενδιαφερόμενοι τα μέτρα, την λήψη αυτών των μέτρων. Και όπως επισημάνατε, όντως το θέμα είναι ιδιαίτερο τεχνικό και γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ακριβείς, ώστε όσοι θα το χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες ε, να μην έχουν προβλήματα, να είναι εύχριστο και ακριβές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι πάντα πρόκληση. Όχι να είναι εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή, αλλά μπορούν και οι ενδιαφερόμενοι να το χρησιμοποιήσουν εύκολα το μέσο αυτό. Επαγγελματίες, δικαστές, δικηγόροι και το καθεξής. Η εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε, που Προενίζεται πολύ αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έδωσε σαφέστατες απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θέσαμε σε αυτό το πρώτο διάλογο. Όντως, θα πρέπει, μια και είναι τεχνικό το θέμα, να είμαστε ακριβείς και σαφείς ώστε να είναι εύχριστο το νομοθετικό μέσο. Αλλά πέραν του τεχνικού χαρακτήρα υπάρχει και θέμα λογοδοσία και διαφάνεια των κοινοτικών πράξεων για να προστατεύσουμε του πολίτε, να προστατεύσουμε τα θύματα και να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρισπέκ. Όντως, μακάρι να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε όλες τις μορφές του εγκλήματος και της, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, χωρίς να ξεχνάμε όμως ταυτόχρονα και τα θύματα. Είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν τους εγκαταλείπουμε στη μοίρα τους ε, για να αντιμετωπίσουν μόνοι τους ε, όλα τα αποτελέσματα αυτών των ε, αδικοπραξιών. Μάλιστα, περνάμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης, αγαπητοί συνάδελφοι που προβλέπει την πρώτη παρουσίαση τριών προτάσεων για το σύστημα πληροφοριών Schengen 2, SIS 2. Χαίρομαι που ο εισηγητής μας, ο κύριος Κοέλιο, είναι παρόν, γιατί αυτός είναι αρμόδιος για δύο από τις προτάσεις που αφορούν το σύστημα πληροφοριών Schengen, κυρίως για τη δικαστική συνεργασία και τον έλεγχο της αστυνομίας και της αστυνομικής συνεργασίας. Ο κύριος Λένερ, που απουσιάζει δυστυχώ σήμερα, αφορά την επιστροφή των παρα, παρατύπως των υπηκών τρίτων χωρών. Ε, θα αντικαταστήσει όμως τον κύριο Λένερ ο κύριος Κοέλιο, που θα μας παρουσιάσει και τα τρία θέματα. Πρώτα όμως θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει μια συλλογική ομαδική παρουσίαση των τριών προτάσεων. Μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή και κατόπιν τους σκιώδεις εισηγητέ για τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Προς το τέλος της συζήτησης θα δώσω το λόγο και στον εκπρόσωπο της Μαλτέζικης Προεδρίας και φυσικά και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δευτερολογήσει και να απαντήσει τις απορίες. Θα ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ρόζενμπεργκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω με το ιστορικό του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν, όπως λειτουργεί σήμερα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και στηρίζει και την αστυνομία και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις και καταπολεμά και την παράνομη μετανάστευση. Το σύστημα περιέχει 72 εκατομμύρια ειδοποιήσεις για άτομα και αντικείμενα. Λειτουργεί σε 29 χώρες και είχε πέρσι 4 δισεκατομμύρια προσβάσεις. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, ένα από τα θεμέλια του συστήματος Σέγγεν και όπως είπα ε, λειτουργεί όλο το 24ωρο. Να σας δώσω κάποια νούμερα. Από όταν ξεκίνησε το ΣΥΣ2 το 2013 και πέρσι, είχαμε πάνω από 37.000 συλλήψεις χάρη στο σύστημα. Ένα στους ε, πάνω από 10.000 άτομα δεν μπόρεσαν να μπουν στην ζώνη Σέγγεν, πάνω από 30.000 αγνοούμενοι βρέθηκαν, πάνω από 150.000 άτομα εντοπίστηκαν για να βοηθήσουν σε ποινικέ διαδικασίες, πάνω από 120.000 ε, εγκληματίες και άλλα άτομα που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια εντοπίστηκαν κτλ. Οπότε τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, το σύστημα λειτουργεί, αλλά ο συνήθως βεβαίως πάντα μπορεί να βελτιωθεί το 2016, τρία χρόνια μετά την έναρξη του ΣΥΣ2, η Κομισιόν έκανε μια αξιολόγηση, όπως απαιτούσε και η νομική βάση, και τα ευρήματα ήταν θετικά, αλλά ε, Βεβαίω υπήρχε και περιθώριο βελτίωσης. Να αναφέρω λοιπόν κάποιους ε, τομείς ε, στους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει βελτίωση. Πρώτα απ' όλα η χρήση από τα κράτη-μέλη, ειδικά οι πληροφορίες ε, στις ειδοποιήσεις ε, και η χρήση των, ε, και η γνώση των χρηστών. Τέλος, η συστηματική αναζήτηση του ΣΥΣ όταν γίνεται αναζήτηση σε εθνική βάση δεδομένων που δεν γίνεται σήμερα. Τέλος, οι ψεύτικες ταυτότητες που θα έπρεπε να διασταυρώνται αυτομάτως με τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ένα άλλο θέμα, οι ελλείψεις ποιότητας δεδομένων, δεδομένα που δεν είναι πλήρη και βάζουν Ένα άλλο θέμα, η δυνατότητα να υπάρχουν οι πόροι, η τεχνική και η λυπη για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αλλαγή του συστήματος πιο γρήγορα. Η ανάγκη να βελτιωθεί η λειτουργική συνέχεια και η διαθεσιμότητα του συστήματος ε, και πάλι και αυτό και τελευταίο οι κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον κανονισμό που θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να επικαιροποιηθεί. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο. Λοιπόν, εάν θέλετε το τεχνικό πλαίσιο, κοιτώντα προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, το πρώτο το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν έχουμε μία πρόταση, αλλά τρεις. Αυτό αντικατοπτρίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με αστυνομική και δικαστική συνεργασία στο ένα μέσο και τους συνοριακούς ελέγχους στο άλλο, αλλά βεβαίως αντικατοπτρίζει και την επιθυμία μας να έχουμε ένα άλλο θέμα το οποίο θα καλύπτεται τις επιστροφές για το οποίο προτείνεται τώρα ένας τρίτος κανονισμός και η τριπλή αυτή δομή είναι αναγκαία, περίπλοκη αλλά αναγκαία, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής των κρατών μελών σε διαφορετικά τμήματα του κεκτημένου Σέγγεν. Οπότε όσο και αν θέλαμε να το αποφύγουμε, η νομική υπηρεσία μας είπε να διατηρηθεί η τριπλή δομή, λόγω της διαφορετικής συμμετοχής των κρατών μελών. Τώρα, να δούμε την ουσία. Πέρα από τις τεχνικές αλλαγές που προκύπτουν ε, απευθείας από την αξιολόγηση, υπάρχουν και κάποιες πιο ουσιαστικές ε, πολιτικές, αν θέλετε, αλλαγές. Ε, η μία αφορά τα βιομετρικά στοιχεία. Αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός των βιομετρικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανταποκριθούμε σε ανάγκε των κρατών μελών. Επίσης, ε, ε, φωτογραφίες ε, προσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα για ταυτοποίηση που επιτρέπει πλέον η τεχνολογία και βεβαίως υπάρχει και βεβαίως η παλάμη, το αποτύπωμα της παλάμης, όπως επίσης και το DNA, το οποίο είναι πολύ σημαντικό βεβαίως όταν έχουμε αγνοούμενα άτομα και δεν υπάρχουν άλλα βιομετρικά δεδομένα. Μία άλλη καινοτομία είναι ότι οι προτάσεις απαιτούν αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων όταν υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα κάποιου, οπότε αν υπάρχει αμφιβολία πρέπει να επαληθεύσουμε το δακτυλικό αποτύπωμα και τέλος οι προτάσεις προβλέπουν μια νέα κατηγορία ειδοποίησης για άγνωστα άτομα τα οποία αναζητούνται σε σχέση με κάποιο έγκλημα και έτσι θα μπορούν να υπάρχουν ειδοποιήσεις για αποτυπώματα δακτυλικά είτε παλάμης όταν ξέρουμε ότι έχουμε το αποτύπωμα ενός δράστη π.χ. σε ένα όπλο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά. Για την αντιτρομοκρατία οι προτάσεις ε, έχουν κάποια μέτρα που στοχεύουν πιο πολύ στην αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα εξής. Πρώτα απ' όλα, υποχρεωτική ε, δημιουργία ειδοποιήσεων για άτομα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Το βασικό εδώ είναι το υποχρεωτική. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα. Δεύτερον, ένδειξη στην ειδοποίηση εάν το άτομο εμπλέκεται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Τρίτον, εισαγωγή μιας νέας ε, δράσης ε, ο λεγόμενος ε, έλεγχος ε, ερώτησης ε, που είναι κάτι μεταξύ του διακριτού ελέγχου και του απλού ελέγχου που έχουμε σήμερα που θα επιτρέπει ακριβώς ένα ενδιάμεσο επίπεδο. Τρίτον, τρίτη κατηγορία λαγών. αφορά τους προληπτικές ειδοποιήσεις. Οι προτάσεις επιφέρουν αλλαγές ειδοποιήσεις για αγνοούμενα άτομα στην περίπτωση στην οποία θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος απαγωγής από γονέα. Και αν γίνει δεκτό σημαίνει ότι εκεί όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος ε, απαγωγής από γονέα ή συνοριοφύλακες και η αστυνομία θα ειδοποιείται και θα μπορούν έτσι να ελέγχουν τις περιπτώσεις τις οποίες ε, ταξιδεύει ένα παιδί και θα παίρνει και το θα μπορεί να κρατεί το παιδί να κρατεί το παιδί για να το προστατεύσει. Τώρα για τις επιστροφές ε, μέσω αυτής της ξεχωριστής πρότασης ε, υπάρχει μια νέα κατηγορία ειδοποιήσεων για άτομα τα οποία δεν έχουν δικαίωμα να παραμπίνουν στην περιοχή Σέγγεν και πρέπει να επαναπατριστούν. Μέσω της εισαγωγής ε, της ειδοποίησης στο ΣΥΣ θα μπορούν ε, οι μεταναστευτικές αρχές ε, να διαπιστώσουν αν τα άτομα αυτά έχουν φύγει από τη ζώνη Σέγγεν και επιπλέον θα ειδοποιούνται οι αρχές όταν τα άτομα αυτά δεν έχουν φύγει. Και έτσι θα μπορέσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιβάλλουν την επιστροφή. Επιπλέον, η εισαγωγή ειδοποιήσεων για τις επιστροφές ε, θα αποθαρρύνει τις δευτερογενείς μετακινήσεις ε, καθώς παράνομοι μετανάστες δεν θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν την ε, επιβολή μιας απόφασης επιστροφής με το να πάνε σε ένα άλλο κράτος μέλος. Δεν θα είναι πλέον υπόθεση ενός κράτος μέλους, θα περνάει ε, σε όλες τις χώρες έγκαιν. Επιπλέον θα ανοίξει τον δρόμο για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνε για τις επιστροφές και τέλος είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το πεδίο εφαρμογή ε, του ΣΥΣ δεν θα αλλάξει με αυτό το νέο μέτρο. Ήδη σήμερα, στην υφιστάμενη νομική βάση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το σύστημα για να ε, στηρίξουμε την λειτουργία της οδηγίας περιπιστροφών και να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Αυτό αφορά και την απαγόρευση εισόδου και την επανείσοδο μέσω των στοιχείων που υπάρχουν στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Μία πέμπτη κατηγορία ουσιαστικών αλλαγών αφορά τους θεσμικούς χρήστες, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα. Και αυτό περιλαμβάνει κύριος ε, τις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Για το Eurojust υπάρχουν τα γνωστά δικαιώματα πρόσβασης. Για την Europol προτείνουμε να επεκταθούν τα δικαιώματα πρόσβασης ε, για να επιτραπεί στην Europol να έχει πρόσβαση σε όλες τις ειδοποιήσεις στο σύστημα και η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό ανταποκρίνεται στην εντολή της Europol όπως αναφέρεται στον κανονισμό και την εμπλοκή της στην καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών και της οξελικής εκμετάλλευσης παιδιών. Τη... Γνωρίζουμε τη σχέση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος και βέβαια υπάρχει ακριβώ αυτό το κενό ενημέρωση, ε, το οποίο θα καλυφθεί μέσω ακριβώς της κοινή εμπειρία για την Frontex ή μάλλον την Ευρωπαϊκή Συνορία Φυλακή και Ακτοφυλακή ε, δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσουν και βεβαίως αυτό σχετίζεται με την ανάγκη διαχείρισης ε, της μετανάστευσης, ε, της λειτουργίας στα hot spot ε, που πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα ΣΥΣ για να υπάρχει ακριβώς κατάλληλη ενίσχυση των κρατών μελών που στηρίζουν. Οι προτάσεις αυτές προβλέπουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, αλλά δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι για τις ειδοποίησεις εκτός εάν τους δώσει την άδεια το κράτος μέλος το οποίο ε, φιλοξενούνται. Θα μπορούν απλά να συμβουλεύονται το σύστημα, αλλά ε, δεν είναι τμήμα της επιβολής. Και βέβαια, η τελευταία υπηρεσία που πρέπει να αναφέρω είναι η Γιουλίζα, η οποία θα παραμείνει αρμόδια για την επιχειρησιακή διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν και αυτό επιβεβαιώνεται από τις προτάσεις, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ειδικά όταν μιλάμε για ποιοτική ανάλυση δεδομένων και στατιστικά στοιχεία που μπορεί να δώσει η υπηρεσία. Και επίσης να υπάρχουν και συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για την Ιουλίζα για συμπληρωματικές πληροφορίες και δοκιμές. Και τέλος, ε, λίγα λόγια για το κόστος. Το συνολικό κόστος ε, για τις επιπρόσθετες αυτές αλλαγές ε, που θα γίνουν ε, από το 18 μέχρι το 2020 προϋπολογίζουμε 67,9 εκατομμύρια ευρώ 64,3 για τεχνική αναβάθμιση για να εφαρμόσουμε τις διατάξεις που αφορούν τα συνοριακά ζητήματα και θα έλεγα το μικρό ποσό των 3,6 εκατομμυρίων, ε, εκατομμυρίων το οποίο αφορά τις επιστροφές και αναγνωρίζουμε βέβαιω ότι θα υπάρχει και κόστος στο εθνικό επίπεδο καθώς απαιτείται η ανάγκη αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων και για τον λόγο αυτόν η Κομισιόν θα διαθέσει 1,2 εκατομμύρια στο κάθε κράτος μέλος ως συνεισφορά που θα γίνει στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης συνόρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι όχι μόνο είναι σημαντικό να συγκεντρώνουμε οποιαδήποτε στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και την ποιότητα αυτών των στοιχείων. Η δεν είναι αποτελεσματική συγκέντρωση απλώς δεδομένων. Ε, θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους πολλαπλούς σκοπούς αυτών των προτάσεων και καλό θα ήταν να έχουμε και προτάσεις περί διαλειτουργικότητας όταν μιλούμε για νέες ιδέες που θα προσθέσουμε στο σύστημα ΣΥΣ. Θα δώσω το λόγο και για τα τρία θέματα στον κύριο Κοέλιο που είναι ο εισηγητής του ΕΛΚ και ένας από τους πλέον πεπειραμένους ευρωβουλευτές για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Κύριε Κοέλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ σφαιρική παρουσίαση και πολύ εμπεριστατωμένη. Όπως ακούσαμε, ε, το ΣΥΣ είναι το σύστημα ε, ε, με τη μεγαλύτερη χρήση. 70 εκατομμύρια ειδοποιήσεις μας είπε ε, για φέτος. 4 ε, δισεκατομμύρια αναζητήσεις είχαμε πέρυσι. Πάνω από 200.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν το 2016, δηλαδή αύξηση 38% σε σχέση με το 2015. Όντως είναι το μεγαλύτερο και πλέον ε, χρησιμοποιούμενο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ε, πληροφοριών σε αφορά το χώρο ασφάλεια ελευθερία και δικαιοσύνη και είναι ε, το σύστημα που αναγνωρίζεται ω μείζον επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη κυκλοφορία, γιατί εξασφαλίζει τα εξωτερικά μα σύνορα και βελτιώνει και την εσωτερική μα ασφάλεια, με και και το βασικό εργαλείο τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ε, έδωσε μάχη για μια διαρθρωμένη, συγκροτημένη ανάπτυξη του ΣΥΣ, ε, φυσικά με σεβασμό των προαναφερθέντων στόχων. Δηλαδή, το σύστημα ΣΥΣ θα πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις ε, αρμόδιες αρχές και φορείς που το χρησιμοποιούν, να εξασφαλίζει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες ε, με ταυτόχρονο σεβασμό και τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν εγκαινιάστηκε το ΣΥΣ2 ζητήσαμε περισσότερες, ε, περισσότερα λειτουργικά στοιχεία, περισσότερες προσβάσεις αλλά και ενδιάμεση αξιολόγηση. Γιατί γνωρίζαμε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΣΥΣ μεταβάλλονται διαρκώς. Αλλά πολλές φορές κάποιες αλλαγές που γίνονται εν θερμό είναι επιζήμιες για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα δεν βελτιώνει κατά πολύ ε, τη διαχείριση των συνόρων ή τη συνεργασία. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ ε, των ε, τριών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Γερούν Λέναρς, που είναι ο εισηγητής για την πρόταση περί επιστροφής, ζητά συγγνώμη γιατί κολλείεται σήμερα. Είναι και αυτός στη Μάλτα, στο συνέδριο του ΕΛΚ. Σε ό,τι αφορά τι επιστροφέ, θα ήθελα να σα πει ότι το ΕΛΚ χαιρετίζει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προσπάθειε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την επιστροφή παρατύπω ε, μεταδιαμενόντων, μεταναστών. Ε, είναι χαμηλό ε, κάτω από 30% ρυθμός επιστροφών με μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων επικοτήτων. Θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό επιστροφών για να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να παρέχουμε προστασία ε, στους πραγματικά χρήζοντες προστασίας. Ε, το σύστημα είναι περίπλοκο. Πέρυσι αντιμετωπίσαμε το θέμα της ενημέρωσης ε, των ταξιδιωτικών εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρούσα πρόταση για την επιβολή της υποχρέωσης στα κράτη-μέλη να εισαγάγουν στο ΣΥΣ σε γραπτές αποφάσεις θα πρέπει να εξεταστεί από αυτό το φως. Πρόκειται για μικρό αλλά απαραίτητο βήμα να αντιμετωπιστεί αυτό το ψηφιδωτό, το περίπλοκο ψηφιδωτό, ε, προκειμένου να μειώσουμε ε, και να αποτρέψουμε τους παράτυπους μετανάστες από το να εισέλθουν στην Ένωση. Επίση, ό,τι αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται στο εφιστάμενο πλαίσιο, ο στόχο είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσει ε, και αυτές που έχουν περιληφθεί στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια. Το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν είναι πολύ ε, ορθολογικό σύστημα και χάρη στις τελευταίες αλλαγές θα βελτιώσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, θα έχουμε περισσότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την ε, αποκαλούμενη προσφυγική κρίση ε, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις επιστροφών θα έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση και συνεργασία των κρατών μελών ε, μεγαλύτερη πρόσβαση στους οργανισμούς που εργάζονται επί τόπου. Επίσης, ε, καλύτερη καταπολέμηση τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος με ανταλλαγή στοιχείων και υποχρέωση έκδοση ειδοποιήσεων για όσου καταζητούνται για τρομοκρατία. Επίσης, θα έχουμε περισσότερα εργαλεία για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Γιατί θα έχουμε ειδικό σύστημα ειδοποίηση για τα παιδιά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Επίσης, η πρόταση ενισχύει την αρχιτεκτονική του συστήματος και προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων, την ασφάλειά τους, την προστασία τους και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη παραπάνω τις προτάσεις αυτές. Καταρχήν, θα πρέπει να έχουμε επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό καλώ του ηγητέ και όδη ηγητέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιε προπαρασκευαστικέ συναντήσει, ώστε να εξετάσουμε διεξοδικά τι επιμέρου προτάσει. Έχω ήδη όμω κάποιε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελα να μου αποσαφηνήσει. Ευθύ εξ αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλωστε ήταν υπέρ του να μην έχουμε εθνικά αντίγραφα, δηλαδή μόνο ένα κεντρικό σύστημα ε, για την έκδοση ειδοποιήσεων και όχι αντίστοιχα αντίγραφα συστημάτων στα κράτη-μέλη. Τότε η επιλογή ήταν να αφήσουμε ε, το θέμα στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Σήμερα και παρά το ότι άλλα συστήματα έχουν κεντρική διαχείριση, όπως το σύστημα εισόδου, εξόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά προτείνει ε, να γίνουν τα εθνικά αντίγραφα υποχρεωτικά για το ΣΥΣ. Ερωτώ λοιπόν, προς τι, γιατί υποβάλλει αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είμαι και πιο σαφής. Ε, ε τι γίνεται, πώς λειτουργήσε το σύστημα το περιορισμένο, για τον ε, προορισμένο χρόνο. Μήπως υπήρξαν κάποια προβλήματα δεν έχουμε επενδύσει αρκετά στο δίκτυο που συνδέει τα κράτη-μέλη με το κεντρικό σύστημα. Υπήρξαν κάποιε αδυναμίε στη λειτουργία του κεντρικού συστήματο και προτείνει τα εθνικά αντίγραφα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, πόσο θα κοστίσει κάτι τέτοιο, γιατί μα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αφιερώσει 1,2 εκατομμύρια, θα χορηγήσει 1,2 εκατομμύρια σε κάθε κράτο μέλο. Μάλλον όμω δεν θα φτάσει αυτό το ποσό. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να επικαιροποιήσουν τα εθνικά του αντίγραφα αν δεν περιλαμβάνουν από σήμερα βιομετρικά στοιχεία. Και τέλος, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως ξέρετε, χθες ενεργοποιήθηκε το άρθρο 50 περί αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. από ό,τι έχω καταλάβει, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσωρινή πρόσβαση στο ΣΥΣ στα θέματα της αστυνομικής συνεργασίας. Τώρα, με την παρούσα κατάσταση και σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να ενταχθεί στο ΣΥΣ για τον έλεγχο των συνόρων. Υπό ποιε προποθέσει θα μπορούσε να το κάνει, Καταρχήν, υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γιατί δεν θα είχε νόημα να ενταχθεί τώρα που φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, να ενταχθεί παρόλα αυτά τελευταία στιγμή στο ΣΥΣ. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο και ευχαριστώ που κάνατε μια σύντομη επισκόπηση και των τριών θεμάτων και που θέσατε και πολύ σαφείς ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για τα τρία θέματα Έχουμε τους ίδιους και οδησίγητες, οπότε θα τους ακούσουμε πρώτα και μετά στους υπόλοιπους, θα ακούσουμε τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Θα ξεκινήσω με, το σκιώδη συγητή, με τη σκιώδη συγήτρια Σοσιαλιστό και Δημοκρατώτη, κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την ε, Κομισιόν που μας παρουσίασε τις ε, προτάσεις και ευχαριστώ ε, τον κύριο Κοέλιο που αναφέρθηκε σε μια σειρά ε, θεμάτων θα ήθελα και εγώ να πω την θέση μας ως σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, καθώς επίσης και τις ανησυχίες μας γιατί συμφωνώ με τον κύριο Κοαγιώ ότι το σύστημα λειτουργεί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί και όντως υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μετά από ε, συνεργασία μεταξύ μας μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει διάλογος με την Κομισιόν αλλά και μεταξύ μας έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να ε, βελτιώσουμε τις τρεις προτάσεις που μας έχουν υποβληθεί. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες καλωσορίζουμε αυτήν την πρόταση της Κομισιόν, ιδιαίτερα τούτη τη στιγμή ε, που πραγματικά πρέπει να δώσουμε στις αρχές μας τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία έτσι ώστε ε, να διασφαλίσουν το επίπεδο ασφάλειας που περιμένουν προς προσδοκούν οι πολίτες μας και που εμείς επιθυμούμε να παράσχουμε στους πολίτες. Ε, είναι μια ε, υποχρέωση που έχουμε εμείς ως νομοθέτες και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε ε, τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικά και να λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο. Δεν ε, πιστεύω ότι υπάρχει άλλο αστυνομικό σύστημα το οποίο να διαχειρίζεται τέτοια ροή πληροφοριών ε, σε πραγματικό χρόνο και με τόσο καλό ε, τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει αυτό το σύστημα και βεβαίως συμφωνούμε να υπάρξει και ειδοποίηση όσον αφορά τρομοκρατικά στοιχεία. Ως σκιώδης ε, πρέπει να, για το θέμα αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι εμείς ως πολιτική ε, ομάδα θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και σωστό να ε, διασφαλίσουμε ότι η αναλογικότητα θα πρέπει να διέπει τα νέα βιομετρικά στοιχεία τα οποία προτείνονται με, το, με τη νέα αυτή πρόταση. Θα πρέπει να υπάρξει διευρυμένη προστασία προστασία ε, των προσωπικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα ε, όσον αφορά το θέμα αυτό των βιομετρικών χαρακτηριστικών που ε, προβλέπει το σύστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει προστασία όλων των συλλεγόμενων δεδομένων και να υπάρχει σωστή διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των πολιτών. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν ε, και επιπλέον ε, ειδοποιήσεις εκτός από όσες ανέφερε ο εισηγητής και για τα θέματα των παιδιών και πρέπει να πω ότι και εγώ η ίδια αλλά και άλλοι συνάδελφοι ζητούμε να υπάρξουν ιδιαίτερες προειδοποιήσεις όσον αφορά παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να απαχθούν από, τους, από έναν από τους δύο γονείς αλλά βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο και σαφές νομικό πλαίσιο ε, ε, όταν έχουμε αγνοούμενους ε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ενηλίκους η αντιμετώπιση από πλευράς των αρχών θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα πρέπει βεβαίως να βοηθηθούν και οι αρχές ώστε έγκαιρα να μπορούν να συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα. Ε, όσον αφορά τώρα την χρήση του ΣΥΣΕ για την επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν ε, παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Εδώ ε, υπάρχουν πολλά ζητήματα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κυρίως ε, εάν, ε, όταν ακούμε την Κομισιόν να λέει ότι δεν θα διευρυνθεί η νομική βάση του ΣΥΣ, αλλά παρόλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί ε, για τις επιστροφές. Πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι αρχές ε, υπεύθυνε για θέματα μετανάστευσης ε, θα πρέπει οπωσδήποτε με σαφή τρόπο να ε, προωθούν τα αιτήματα. Συμφωνούμε με κάποιους προβληματισμούς του εισηγητού όσον αφορά τον, την χρηματοδότηση και η Κομισιόν μας είπε ότι 68 εκατομμύρια περίπου θα δοθούν μέχρι το 2020 αλλά δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το τι θα γίνει μετά από την ημερομηνία αυτή ε, θα είναι αυτοστηριζόμενο. Το σύστημα προβλέπει κάτι άλλο η Κομισιόν. Όσον αφορά ας πούμε την πρόταση για τους ε, ε, ελέγχους των ε, συνόρων ε, προτείνεται ότι θα χρηματοδοτηθεί από το σύστημα εσωτερικής, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αλλά δεν αναφέρεται τι θα γίνει με το σύστημα εισόδων-εξόδων όταν θα συνεχιστεί το σύστημα αυτό. Επίσης ε, η Κομισιόν λέει ότι εάν έχει συλλεγεί ε, ένα συγκεκριμένο αριθμός δεδομένων, τότε το άτομο έχει δυνατότητα να ζητήσει πρόσβαση ε, στα στοιχεία αυτά. Θα θέλαμε να μας πει η Κομισιόν κάποια επιπλέον στοιχεία όσον αφορά το θέμα αυτό. Επίσης έγινε αναφορά σε... Fingerprints σε άγνωστους ε, καταζητούμενους ε, ε, θα πρέπει να δούμε τι είδους αδικήματα καλύπτονται όταν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και πώς μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργήσει αυτό. Και κάτι τελευταίο ε, σχετικά ε, με το ότι το, ε, το, το κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για αποζημίωση εάν ζημιωθεί κάποιος πολίτης. Τι είδους ζημία, μιλάμε για οικονομική, για φυσική. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μίριαμ, λέει η Πρόεδρος. Πολλά ερωτήματα, τα οποία θα απαντήσει μάλλον η Κομισιόν αργότερα. Ο κύριος Άλλα από την ECR. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ECR αναγνωρίζει τα προβλήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση και το έγκλημα και την ε, επιτακτική ανάγκη να βρεθούν λύσει στα προβλήματα. Είμαστε υπέρ των στόχων της πρότασης ε, και ε, υπέρ των περισσότερων προτάσεων. Δεν πρόκειται να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειε. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση και ένα σχόλιο. Εν μέρη το κάλυψε ο κύριος Κοέλιο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι πέραν του κεντρικού ΣΥΣ, το σύστημα περιλαμβάνει και εθνικές ε, συνιστώσεις. Δηλαδή κάθε χώρα θα πρέπει να θεσπίσει μερικό ή πλήρως, πλήρες αντίγραφο του συστήματος ΣΥΣ ε, και ένα σύστημα ε, backup. Θεωρώ βέβαια ότι οι κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν για το τι τεχνική λύση θα χρησιμοποιήσουν ε, προκειμένου να εφαρμόσουν τον κανονισμό για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν θέλουν να, ε, να θέσουν ερωτήματα απευθεία στο κεντρικό ΣΥΣ ή να δημιουργήσουν εθνικό του αντίγραφο τη βάση, θα πρέπει να ε, εναπόκειται στην κρίση του. Όταν θεσπίστηκε πριν από λίγα χρόνια το ΣΥΣ 2, τα κράτη-μέλη αποθαρρύνθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουν εθνικό αντίγραφο ενός αρχείου με δεδομένα, αλλά να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και τα αιτήματά του για παροχή πληροφοριών απευθεία στο κεντρικό ΣΥΣ. Η θέσπιση εθνικών αντιγράφων ΣΥΣ για με backup δεν θα είναι αποτελεσματική οικονομικά λύση για να λύσει τα προβλήματα πρόσβασιμότητας. Αρκεί να είναι το κεντρικό ΣΥΣ και το backup που θα έχει αρκετά αποτελεσματικά. Επίσης, με εθνικά αντίγραφα θα είναι πιο ευάλωτο το σύστημα και πιο εκτεθειμένο σε διαρροές. Θα πρέπει να δούμε τις δύο πτυχές του βασικού συστήματος και του συστήματος στήριξης του επικουρικού του backup. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα και οι δύο πλευρές να λειτουργούν ταυτόχρονα. Πέραν όμως ε, ε, αυτού του σημείου της μικρής επιφύλαξης, ε, γενικώ η ομάδα συντηρητικών μεταρρυθμιστών είναι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Χαλάχο. Ο κύριος Δεπρέ είναι ο τελευταίος και ο από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που πολύ εύστοχα ε, είπαν οι προλαλήσαντες για το ΣΥΣ και τις γενικές παρατηρήσεις ε, του εισηγητού για το ΣΥΣ. Δεύτερον, δεν είχα ακόμη αρκετό χρόνο για να διαβάσω διεξοδικά και ενδελεχώ τι τεχνικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σταθώ όμω σε τρία προβλήματα που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πρόβλημα τη ενίσχυσης και τη συμπεριλήψή ε, ε, του ΣΥΣ ε, πέραν των δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών του προσώπου. Κατάλαβα καλά ότι τα κράτη-μέλη που έχουν και τέτοια δακτυλικά αποτυπώματα παλάμης ή φωτογραφίες προσώπου δεν είναι υποχρεωμένα να τα εντάξουν αυτά τα στοιχεία στο ΣΥΣ. Δίνανται, αλλά δεν ε, οφείλουν. Για παράδειγμα, αν έχουμε στοιχεία για έναν τρομοκράτη ε, υποπτώ τρομοκρατίας ε, που με ε, πλαστή ταυτότητα φεύγει από το κράτος ε, που έχει τέτοια στοιχεία, φωτογραφία και ούτω καθεξής. Αυτό συνέβη. Πολλοί χρησιμοποίησαν πλαστές ταυτότητες για να μπουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αν δεν υπάρχει υποχρέωση μετάδοσης αυτών των πληροφοριών θα κυκλοφορούν πολύ πιο εύκολα οι εγκληματίες. Ε, πολύ πιο εύκολα από άλλους που έχουν περιληφθεί στο σύστημα για άλλους λόγους. Είναι δυνατόν ένα κράτος που διαθέτει αυτά τα στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώματα, παλάς ή προσώπου για υπόπτους τρομοκρατίες ή για καταδικαστέντες για εγκλήματα τρομοκρατίες, να μην είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη αυτών των στοιχείων στο κεντρικό ΣΥΣ, αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά κάποιες θετικές απαντήσεις, τη παροχής πληροφοριών, κάποια hits, που αφορούν τρομοκράτες δεν θα πρέπει αυτά αυτόματα να μεταβιβάζονται στην Ευρωπόλ, γιατί η Ευρωπόλ έχει ειδικό τμήμα κατά πολέμηση της τροποκρατίας. Αν δεν έχει όλα τα στοιχεία η Ευρωπόλ, πώς θα επιτελέσει το έργο της για να κάνει την ανάλυση, την επεξεργασία και να το διαθέτει στα κράτη-μέλη. Γιατί να μην προβλέψουμε κάθε φορά που έχουμε, μια συγκεκριτική έτσι παροχής πληροφοριών για πέρασμα και από αστυνομικό έλεγχο, να μεταδίδεται αυτό το hit κατευθείαν στην Ευρωπόλ για να επιτελέσει το έργο της σωστά. Σε ό,τι αφορά τις ε, αρνήσεις ε, εισόδου και διαμονής. Αν κατάλαβα καλά, αυτή τη στιγμή ένα κράτος μέλος δύναται να περιλάβει στο ΣΥΣ μια ειδοποίηση κάποιους για τον οποίο έχει το αίτημα εισόδου. Με τη νέα πρόταση θα ζητήσουμε να συμπεριληφθεί ένδειξη στο ΣΥΣ κάθε φορά που απορρίφθηκε το αίτημα εισόδου με βάση την οδηγία του 2008. Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, εξεκολουθεί να είναι προαιρετικό αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Για παράδειγμα, έχουμε κάποιον ε, που κηρύσσει μυσαλόδοξα ε, θέματα και που επιστρέφει στη χώρα του για την οποία ε, για αυτόν τον άνθρωπο ε, προβλέπεται από το Βέλγιο πενταετής, πενταετής απαγόρευση εισόδου. Αλλά δεν το κοινοποιεί. Θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος ε, ε, που είναι κήρυκας ε, μίσους να, να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια από άλλο κράτος, αφού το Βέλγιο δεν έχει κάνει την κοινοποίηση για την απόρριψη εισόδου. Αν δεν έχουμε συστηματική ειδοποίηση ε, ειδικά σε θέματα που χρειάζονται, όπως είναι η καταπολέμηση των πραγματικών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας, ενώ το έχουμε για άλλους λόγους, τι να πω. Γιατί να μην έχουμε αυτόματη κοινοποίηση σε περίπτωση σοβαρής εγκληματικότητας ή τρομοκρατίας. Αυτά. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως μία απάντηση είναι ότι έχουμε τόσες πολλές βάσεις δεδομένων για τόσους σκοπούς που δεν ξέρω αν η λειτουργικότητα θα βοηθήσει. Ίσως η Κομισιόν να έχει κάποιες πρώτες απαντήσεις, αλλά πριν επανέλθω στην ε, Κομισιόν ε, και τον εισηγητή, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Προεδρία του Συμβουλίου και ελπίζω η εκπρόσωπος να μας ε, πει πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Έχετε τον λόγο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνούμε πως το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της Ευρώπης και έχουμε μια ευθύνη να προχωρήσουμε το θέμα αυτό για το μέλλον της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για μια προτεραιότητα της Μαλτεζικής Προεδρίας και έχουμε συγκαλέσει επιπλέον συναντήσεις για να προχωρήσουν οι συζητήσεις. Μία λεπτομερής εξαγωγή ένα άρθρο των τριών προτάσεων γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα εργασίας ε, και εκτιμένου σε Η Προεδρία σκοπεύει να ολοκληρώσει την πρώτη εξέταση και των τριών προτάσεων μέχρι το τέλος του Μαΐου. Και βεβαίως θέλουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και να δώσουμε οποιαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία. Όμως, ε, με χαρά σημειώνουμε ε, και καλό είναι να σημειώσετε ότι η φάση του τριμερούς διαλόγου θα γίνει επί Εσθονικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Κομισιόν και αν θέλετε και αν μπορείτε βεβαίως να απαντήσετε στις ερωτήσεις, παρακαλώ απαντήστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Κοέλιο και τους κοιόδης εισηγητές που παρουσίασαν τις πρώτες τους ε, παρατηρήσεις. Λοιπόν, ε, καλωσορίζω την πρώτη πρόταση του κυρίου Κοέλιο να ε, γίνουν τεχνικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις, να πάμε σε κάποια από αυτά τα ζητήματα εις βάθος, γιατί βεβαίως είναι τεχνικό το θέμα και απαιτείται περισσότερος χρόνος να συζητηθούν κάποια ζητήματα, γι' αυτό επιμένουμε. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Κοέλιο, ο οποίος όπως αναφέρατε είναι ένας από αυτούς ε, τους αιθούσεις που γνωρίζουν καλύτερα το σύστημα. Θα έλεγα πως από τη δική μας Σκοπιά είναι ε, ένας εκ των ιδρυτών του συστήματος. Χαιρόμαστε λοιπόν που αποδέχτηκε ξανά την ε, ευθύνη για να καταρτήσει την θέση του Κοινοβουλίου για τις νέες αυτές προτάσεις και τον ευχαριστούμε. Για τις ερωτήσεις σας λοιπόν, γιατί ε, προτείνουμε εθνικά αντίγραφα. Το έθεσε και ο κύριος ε, Χαλοάλο. Ε, α, είναι και για μας ε, πονοκέφαλος και το σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά έχετε απόλυτο δίκιο ότι ε, Βεβαίω ω θέμα αρχής ε, μια κεντρική λύση θα ήταν προτιμητέα αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα το SIS είναι ένα υβριδικό σύστημα δηλαδή το πώ έχει εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου και έχει γίνει ένα επιτυχημένο σύστημα που λειτουργεί, αυτό έγινε βασιζόμενο στην μεικτή αρχιτεκτονική, ένα κεντρικό σύστημα δηλαδή το οποίο στηρίζουν εθνικά συστήματα και έχουμε σήμερα 24 κατημέλη που έχουν ένα εθνικό αντίγραφο, μόνο 5 δεν έχουν. Και στις επαφές μας με αυτά τα κράτη-μέλη μάθαμε πως πολλές από τις χώρες που έχουν εθνικό αντίγραφο το εκτιμούν, έχουν επενδύσει σε αυτό και δεν θα ήθελαν να χάσουν αυτή τη δυνατότητα. Υπόθηκε και σωστά ότι το σύστημα δεν έχει πέσει τα τελευταία χρόνια. Πάντα λειτουργούσε το κεντρικό σύστημα, αλλά μπορούμε να πούμε και το αντίστροφο ότι λειτουργούσε γιατί ε, το στήριζαν 24 εθνικά αντίγραφα που βεβαίως ε, έπαιρναν ε, μεγάλο κομμάτι αυτής της κίνησης, της κυκλοφορίας που υπάρχει όλο το 24ωρο στο σύστημα. Μην ξεχνάτε επίσης ότι όταν συζητήσαμε το SIS πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχαν πράγματα όπως η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας. Τα 4 εκατομμύρια ερωτήματα που λαμβάνουν χώρα σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με αυτόματες αναζητήσεις που απαιτούν άμεσες απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να δοθούν ακριβώς λόγω της υβριδικής ε, αυτής αρχιτεκτονικής. Βεβαίως ε, και υπάρχει και χρήση στα σύνορα που πλέον θα είναι συστηματική θα έχουμε συστηματικό έλεγχο του κάθε ταξιδιώτη στα εξωτερικά σύνορα και πάλι στα πραγματική ζωή οι σύνοριοφύλακες δεν θέλουν να περιμένουν οπότε οποιαδήποτε τεχνική λύση μπορεί να στηρίξει την αξιοπιστία του συστήματος ε, και να μειώσει την ευπάθεια ε, είναι θετική. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο καταλήξαμε σε αυτή την σύσταση, αλλά βεβαίως είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω συζητήσεις ε, και με εσά, αλλά και στο Συμβούλιο που ετέθη το ζήτημα. Η δεύτερη ερώτησή σας αφορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ενεργός χρηστής ε, του SIS στο θέμα της αστυνομικής συνεργασίας Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα το θα γίνει σε δύο χρόνια όπως και με όλα τα άλλα θέματα δεν ξέρουμε. Είναι ανοιχτό το ζήτημα για όλους. Για κάποια από τα άλλα ζητήματα δεν θα μπω στα τεχνικά θέματα γιατί είναι καλύτερο να το συζητήσουμε κάπου αλλού αλλά ε, για την προστασία δεδομένων που ανέφερε η κυρία Νταλή πράγματι πάρα πολύ σημαντικό θέμα θεωρούμε, πιστεύουμε ότι οι προτάσεις που ενέκρινε η Κομισιόν αντικατοπτρίζουν ε, τους τελευταίους κανόνες που υπάρχουν για την προστασία των δεδομένων κάναν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ε, π.χ. για κανόνες διαγραφής δεδομένων για απαιτήσει αναλογικότητας ε, όταν θέλουν να επεκτείνουν τα κράτη-μέλη την ημερομηνία λήξης κανόνες αναφοράς ε, συμβάντων, ε, μικρότερες περίοδους διατήρησης ε, αντικειμένων, π.χ. αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και πολύ σαφείς όροι για τη χρήση βιομετρικών δεδομένων. Οπότε θεωρούμε ότι ε, είναι πολύ σύγχρονες οι προτάσεις, αλλά βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Χρηματοδότηση μετά το 2020. Η εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι βεβαίως από εσά εξαρτάται, δεν θα το αποφασίσει η Κομισιόν. Αλλά νομίζω μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι ένα σύστημα απαραίτητο που λειτουργεί πάντα θα ε, βρει τρόπους ε, να χρηματοδοτηθεί. Οπότε, ε, μας περιπτώσει θα είναι προτεραιότητα για εμάς ε, Βεβαίω ε, οι προτάσεις αυτές ε, για τα έξυπνα σύνορα είχε, είχαν οργανωθεί και συζητηθεί και εδώ μέσα νομίζω και βεβαίως ε, μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικές οικονομίες στο θέμα των έξυπνων συνόρων που είχαν αρχικά πολύ υψηλότερο προϋπολογισμό όπως φάνηκε ε, μετά τις ε, δοκιμές μας ε, που κατέληξαν στην πρόταση για το σχετικό σύστημα τον Απρίλιο πέρσι. Από εκεί λοιπόν είναι τα χρήματα για την ευθύνη των κρατών μελών. Για... Είναι σε όλες τις κατηγορίες, δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για κάθε πτυχή, για... είναι... έχουν αστική ευθύνη για κάθε πτυχή που είναι υπεύθυνα. κάτι τελευταίο για αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Ντεπρέ. Για τα βιομετρικά δεδομένα η κατάσταση σήμερα είναι ότι υπάρχει υποχρέωση να ανεβαίνουν τέτοια δεδομένα όπου αυτό έχει σημασία αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση να χρησιμοποιούνται. Και αυτό είναι το νέο στοιχείο. είναι φανταστικό να γεμίζουμε το σύστημα αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε κιόλας. Αυτό είναι το νόημα. Σήμερα βλέπουμε συχνά ότι τα κράτη-μέλη για οποιονδήποτε λόγο και φαντάζομαι ότι πολλοί από αυτούς τους λόγους είναι θέμητοι δεν ε, αναζητούν ε, σε όλες τις καταστάσεις που έπρεπε. Αυτό σκοπεύει λοιπόν να κάνει. Και σκοπεύει να κάνει την διαφορά η πρόταση για την Europol. θα έχει μεγαλύτερο ρόλο. Τώρα, αν θα είναι υποχρεωτικό η Europol να δίνει αυτές τις πληροφορίες σε όλους, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι δυνατόν. Αυτό αφορά το ποιο έχει την ειδοποίηση. Δηλαδή, η Europol ε, φιλοξενεί, αλλά δεν είναι ο κάτοχος αυτών των δεδομένων. Κάτοχοι είναι τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα έχει πρόσβαση και για την απαγόρευση εισόδου, το τελευταίο το οποίο είπατε. Σήμερα είναι ήδη υποχρεωτικό να μπαίνει στο SIS, να μπαίνουν οι απαγορεύσει εισόδου που αφορούν ε, τα σοβαρά εγκλήματα και την τρομοκρατία, αλλά όχι ακόμα για την μετανάστευση. Οπότε, εάν βρεθεί μια απόφαση επιστροφής ε, και υπάρχει και απαγόρευση εισόδου από το κράτο μέλο που την εξέδωσε, δεν υπάρχει υποχρέωση, δεν υπάρχει δυνατότητα, δυνατότητα υπάρχει, δεν υπάρχει υποχρέωση να μπει στο σύστημα. Το, αυτό θα είναι το νέο στοιχείο για να ε, λειτουργεί το SAS και στον τομέα των επιστροφών. Νομίζω ότι κάλυψα κάποιες, ερω... κάποιες ερωτήσεις, όχι όλες, ε, αλλά είμαι στην διάθεσή σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως ε, ε, μας δώσατε πολλές πληροφορίες. Θα ζητήσουμε και επιπλέον πληροφορίες στη διάρκεια της διαδικασίας ε, και για θέματα βεβαίως τα οποία σχετίζονται με τα εθνικά αντίγραφα και το, τι, τι, τι θα γίνει με αυτά θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κοέλιο, τον εισηγητή, για κάποιες ε, τελευταίες ε, ε, παρατηρήσεις. Ναι, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις και για το input. Ευχαριστώ βεβαίως και την Κομισιόν η οποία είναι διατεθειμένη να μας συνδράμει ε, στη διάρκεια της τεχνικής διαδικασίας. Ε, νομίζω ότι μπορώ να πω και εγώ ότι η ασφάλεια είναι βασική ε, αξία και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πολίτες μας. Και νομίζω ότι και οι σκιώδεις συμφωνούν ότι μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συμφωνία στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοέγελε, η Πρόεδρος. Ε, να πω ότι οι δύο εισηγητές θα υποβάλουν προσχέδια έκθεσης στην ε, Επιτροπή μας ε, ΛΥΜΠΕ τον Ιούνιο. Επομένως, η απόφαση όντως θα ληφθεί υπό Εστονική Προεδρία με τις καλύτερες συνθήκες να σας πω ότι το επόμενο θέμα ξεκινάει στις 11.45, ε, οπότε μπορείτε να βγείτε, να πιείτε νερό, να πιείτε καφέ, να ξεκουραστείτε λίγο, αλλά οπωσδήποτε να είστε εδώ 11.45, προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του επόμενου θέματος.

Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρος, θα συνεχίσουμε τώρα την συνεδρίασή μας, την πρωινή μας συνεδρίαση, καλωσορίζοντας θερμά ε, την κυρία ε, Μπονίτσι, ε, ε, η οποία είναι πρέσβη στη μόνιμη προσωπία της Μάλτας ίσα την στις ε, ε, Βρυξέλλες ε, και θα ήρθε εδώ έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τα συμπεράσματα και για τα τεκτενόμενα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχετε 10 λεπτά για θεωρητικός, αλλά βεβαίως με την ησυχία σας μπορείτε να μας τα πείτε όλα αυτά που θέλετε και μετά ε, θα ξεκινήσει η συζήτηση. Κύρια Μπονίτζη, έχετε το λόγο παρακαλώ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Όπως ξέρετε, στην αρχή της εβδομάδος ε, είχαμε το Συμβούλιο ΔΕΗ την Δευτέρα 27 Μαρτίου ε, οι εσωτερικές υποθέσεις ε, υπό τον αρμόδιο Υπουργό Καρμέλο Αντένα και τα θέματα δικαιοσύνης την 28 Μαρτίου υπό την ε, Προεδρία της ε, κυρίας ε, Μπονίτσι, αρμοδίας Υπουργού. Στα δύο και στα δύο τμήματα αναφερθήκαμε στα τραγικά περιστατικά που συνέβησαν στο Λονδίνο την προηγούμενη εβδομάδα που μας ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο την πεποίθηση ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Ε, βεβαίως ε, θυμηθήκαμε και τα τραγικά περιστατικά που έλαβαν χώρα στο Βέλγιο ένα χρόνο πριν. πρέπει να προσπαθήσουμε να προλάβουμε στο μέλλον όσο γίνεται περισσότερο τέτοιου είδους περιστατικά έτσι ώστε οι πολίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς. Μετά ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα, μελετούμε τα θέματα εσωτερικών υποθέσεων και ασχοληθήκαμε με τα ε, θέματα με τη σειρά που σας αναφέρω. Ε, πρώτα απ' όλα ε, αναφερθήκαμε στο θέμα το μεταναστευτικό σύμφωνα με τα συμπεράσματα της την δήλωση της Μάλτας του Φεβρουαρίου 2017. Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερως με τους διαδρόμους των μεταναστευτικών ροών και ε, προσπαθήσαμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική ε, εφαρμογή της δήλωσης της Μάλτας. Δυστυχώς ε, φαίνεται ότι ακόμα είναι υπερβολικά πολλοί οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στην Μεσόγειο και έρχεται η Άνοιξη και φοβούμαστε ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε ε, να εργαζόμαστε μαζί με τους διεθνείς μας εταίρους, πάντα με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι αυτονόητο φυσικά. οι δράσεις οι οποίες αναφέρονται σε τη δήλωση της ε, Μάλτας και που μεταφράζονται και αντικατοπτρίζονται και στο σχέδιο δράσης ε, καταδεικνύουν ότι έχουν ε, καταβληθεί όλες οι σχετικές προσπάθειες. Αυτό σημαίνει οικοδόμηση ικανοτήτων όσον αφορά την ακτοφυλακή, βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των μεταναστών στους καταβλισμούς, και ε, καταπολέμηση των εγκληματικών ε, ομάδων, βοήθεια στην εθελούσια επιστροφή, ε, δυνατότητα εξέβρεσης εναλλακτικών μορφών για εισόδημα έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτή η ε, υποβοήθηση ας πούμε της ε, παράτυπης ε, μετανάστευσης. Φυσικά οι δυσκολίες υπάρχουν και παραμένουν και πολλές δυσκολίες απορρέουν από την κατάσταση στην Λιβύη. Δεν θέλουμε να είμαστε αφελείς και πρέπει παρόλα αυτά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ε, στο Συμβούλιο ε, Εσωτερικών Υποθέσεων επίσης ε, υπήρξε μια ενημέρωση για το σχέδιο δράσης της Βαλέτα, απόρρια της διάσκεψης της Βαλέτα του 2015 στην ε, ε, Μάλτα πριν από, από ένα μήνα ε, έλαβε χώρα και μια άλλη συνεδρίαση για την συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου δράσης της Βαλέτα. Επίσης, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι οδήγηθηκαν σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία τώρα θα πρέπει να υλοποιηθούν βάσει και των διαδικασιών της Χαρτούμ και θα συζητηθούν ε, περαιτέρω ε, το πρώτο τρίμηνο του 2018 στη διάσκεψη την οποία, η οποία θα ε, λάβει χώρα στην Αιθιοπία. Επίσης συζητήθηκε η υλοποίηση της επαναπρόθεσης And συγγνώμη, της μετεγκατάστασης ε, έτσι ώστε να καταβληθούν όλες ε, οι προσπάθειες ε, και αυτές να καταβληθούν έγκαιρα. Επίσης, είναι θεμελιώδου σημασία να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί, διότι η Ιταλία και η Ελλάδα εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να υλοποιηθούν οι συμφωνίες. Όσον αφορά την πολιτική επιστροφών, ε, έγινε συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών ε, πάνω στην ανακοίνωση της Κομισιόν των αρχών Μαρτίου. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικότερης πολιτικής επιστροφών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ε, δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, κυρίως σε δύο στοιχεία επικεντρώθηκε η συζήτηση. Ε, η συνεργασία ε, με τις τρίτες χώρες, αλλά και σε επίπεδο να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κατάχρηση των συστημάτων επιστροφών από τα κράτη-μέλη. Ε, η μεταρρύθμιση του συστήματος ε, ΣΥΙΣΕ επίσης είχε εγγραφεί στη μέσα Διάταξη ε, και παρουσιάστηκε, υπευλήθη στους υπουργούς μια έκθεση πρόοδου. Ε, το θέμα αυτό, η δέσμη αυτή είναι υψηλή ε, προτεραιότητα, Επίσης, ε, ο κανονισμός του Δουβλίνου, έτσι όπως συζητήθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Εμεί έχουμε συνεχίσει τις διαδικασίες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, έτσι ώστε να επιτύχουμε την ε, επαρκή και αποτελεσματική υλοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης. Ε, επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου έχει ξεκινήσει διαδικασίες και διαβουλεύσει με το Κοινοβούλιο και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία. Βεβαίως η υπηρεσία ασύλου θα εξακολουθήσει να ε, λαμβάνει και να διεκπεραιώνει όσες περισσότερες αιτήσει ε, μπορεί. Ε, επίσης η διαχείριση των συνόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Με χαρά βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις όσον αφορά το σύστημα αίτηση και ευελπιστούμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε περισσότερες ε, περισσότερα στοιχεία. Όσον αφορά τα θέματα δικαιοσύνης ε, που όπως σας είπα συζητήθηκαν την επόμενη μέρα στις 28 Μαρτίου. Συζητήθηκαν αρκετά θέματα μεταξύ των οποίων αυτά που σας αναφέρω τώρα. Σε ό,τι αφορά την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, οι Υπουργοί Δικαιοσύνη ε, άκουσαν την έκθεση πρόοδο για την κατάσταση και με βάση τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και τα περσινά αποτελέσματα α, συζητήθηκαν διάφορες πτυχές του θέματος σε τεχνικές συζητήσεις. Σημειώθηκε πρόοδος σε, φορά, σε πολλά θέματα όπως κριτήρια συμμόρφωσης, κανόνες για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου υπηρεσιών και σε περίπτωση μη τήρησης υπηρεσίες ποιες δυνατότητες μέσων υπάρχουν για την αποκατάσταση. Επίσης, ε, με τα μέτρα αυτά πιστεύουμε θα έχουμε μεγαλύτερη πρόοδο προς την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ε, Ενίας Ψηφιακής Αγοράς προς το συμφέρον κυρίως των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Καταρχήν, κα, τα εμπόδια από ε, το σχετικό δίκτυο. Επίσης, έρονται τα εμπόδια που οφείλονται στις διαφορές μεταξύ του ενοχικού δικαίου των χωρών μελών. Θα υποφεληθούν έτσι οι επιχειρήσει και οι καταναλωτέ και από αυτού. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του διεθνού εγκλήματο και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, οι ε, υπουργοί άκουσαν έκθεση πρόοδου για την πρόταση οδηγία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη νομοποίηση όδων από παράνομε δραστηριότητε, ποινικού δικαίου και επίση τα θέματα βιβαία αναγνώριση των ανταλμάτων δέσμευση και δίμευση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του σχεδίου δράση για την αναβάθμιση και ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας επίσης εξακολουθεί να συνιστά η προτεραιότητα, όπως η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητα για τους πολίτες. Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος ε, στην πρόταση της αντιμετώπισης του ξεπλήματος χρήματος από το ποινικό δίκαιο και η πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση των ενταλμάτων δέσμευσης και δίμευσης είναι ένα πιο περίπλοκο, εκτενέστερο και πιο ουσιαστικό νομοθέτημα, γι' αυτό θα απαιτήσει ε, μια πιο χρονοβόρα διαδικασία εξέτασης. Πάντω και οι δύο προτάσεις θα μα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία από πολλέ πτυχέ, εξασφαλίζοντα τα απαραίτητα μέσα και μηχανισμού στα κράτη-μέλη, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτέ τι νέε απειλέ που προέρχονται από τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Ένα άλλο θέμα στο πρόγραμμα του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη ήταν η επιστροφή των ξένων ε, τζιχαντιστών. Ένα άλλο μείζον πρόβλημα που αντιμετώπισαν πολλές χώρες μέλη. Οι υπουργοί συζήτησαν κάποια μέτρα πολιτικής ε, που υπέβαλε ε, το Συντοριστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας προκειμένου να, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου. Στο δείπνο, οι υπουργοί συζήτησαν το θέμα των καταγγελόντων και της ενίσχυσης προστασίας των καταγγελόντων, γιατί οι καταγγέλοντες ε, ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δημοκρατικές κοινωνίες, ε, αποκαλύπτοντας αθέμητη παράνομη συμπεριφορά για θέματα δωροδοκίας, απάτης, χρηματισμού και του καθεξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε τη δική του έκθεση για το θέμα αυτό της προστασίας των καταγγελόντων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσιες διαβουλεύσεις. σκοπός της συζήτησης στο δείπνο ε, ήταν να δοθεί μια ευκαιρία στους Υπουργούς Δικαιοσύνης να ανταλλάξουν ε, απόψεις για το θέμα αυτό. Και τέλος, ό,τι αφορά ε, τις άτυπες συζητήσεις που έγιναν για το σχέδιο κανονισμού για την ε, σύσταση του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό έγινε στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης. Όπως θα θυμάστε, στις αρχές του μήνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε αυτό το θέμα και άνοιξε το δρόμο για ενισχυμένη συνεργασία προκειμένου να ιδρυθεί η, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Πάντως η συνάντηση αυτή δεν έγινε στα πλαίσια του επίσημου συμβουλίου, μια και το σχέδιο κανονισμού έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Έχει, έχουν διακοπεί σχετικέ συζητήσεις. Έγινε στο πλαίσιο μια άτυπη συνάντηση που διευκόλυνε η Μαλτέζικη Προεδρία. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειε για το θέμα τη Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή. Πάντω, η άτυπη αυτή συζήτηση που έγινε την Τρίτη έδωσε την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως οι Υπουργοί για τα επόμενα βήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερο συντονισμό. Η Προεδρία πάντως θα συνεχίσει να ε, παρέχει χώρο συζήτησης για τις μελλοντικέ συζητήσεις. Και... ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες για ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών και να σας υπενθυμίσω παρά το ότι είμαστε στη ΛΥΜΠΕ ότι βεβαίως όταν μιλάμε για την ασφάλεια και τη μετανάστευση υπάρχει και μια εξωτερική διάσταση που πρέπει να μας απασχολήσει για να βρούμε μια λύση και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις εσωτερικές μας δυνατότητες. Αλλά βεβαίως εδώ στην Λίμπε μιλάμε για τις εσωτερικές μας δυνατότητες, γι' αυτό έχουμε και εκπροσώπους από την Κομισιόν, την Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης ε, και Εσωτερικών και θα δώσω λίγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Φωνσέκα Μαρία για να προσθέσει κάτι για τα θέματα δικαιοσύνης. Κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Μπονίτσι, κυρίες και κύριοι, μετά την ε, ε εξαντλητική ενημέρωση που μας έκανε η πρέσβη Μπονίτσι, δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Απλώς, ε, ξεκινώντας από την ερώτησή σας, να επιβεβαιώσω ότι οι άτυπε συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έγιναν και οι διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές ε, για ένα τόσο περίπλοκο θέμα που άπτεται το άρθρο 86 της συνθήκης. Θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς στην πρόθεση της συζήτησης προκειμένου να καταλήξουμε σε αίσιο αποτέλεσμα. Βέβαια, στην καλύτερη περίπτωση οι επίσημες συζητήσεις θα αρχίσουν ε, την επόμενη εβδομάδα. Θα εξαρτηθεί από το θα, αν θα έχουν υπογράψει τη σχετική επιστολή τα κράτη-μέλη. Εμείς είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη, θα ήθελα και εδώ να σας επιβεβαιώσω ότι στην συζήτηση ανατολισμού που έγινε για την ε, ποινική δικαιοσύνη και την ε, αντίδραση ποινική δικαιοσύνη στον κυβερνοχώρο. Ήταν μια σφαιρική συζήτηση, εξαντλητική. Τρεις υπουργοί μίλησαν πολύ ανοιχτά για την, ε, για την συνοχή, το... τη συνάφεια των θεμάτων, προστασία των δεδομένων, ηλεκτρονικές ταυτότητες, κρυπτογράφηση, κωδικοποίηση Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τις προθεσμίες και θα υποβάλει εγκαίρως την έκθεσή της μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο του Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά τα τις ψηφιακές συμβάσεις, περιμένουμε τη γενική θέση του Συμβουλίου τον Ιούνιο υπό την αιγυδά της Προεδρίας και πιστεύουμε ότι και για το θέμα αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε έναν αυστηρό παραλληλισμό και εξισορρόπηση μεταξύ αφενός των αναγκών των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά αλλά και της προστασίας των καταναλωτών που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αλλά περιμένουμε να συνεχιστούν οι συζητήσεις ώστε να καταλήξουμε σε αυτή τη γενική άποψη, γενική προσέγγιση του Συμβουλίου τον Ιούνιο για τους ε, καταγγέλλοντες επιβεβαιώνω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ύψιστη πολιτική σημασία που έχει αυτό το θέμα και αναζητεί την πιο συνεκτική προσέγγιση προκειμένου σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να υποβάλει τις προτάσεις της ε, εν ευθέτω χρόνο και εμπρόθεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την μελλοντική συνεργασία λοιπόν με το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μας τελευταίους μήνες και χρόνια έχει επιδείξει ότι αν είναι αναγκαίο εμείς εργαζόμαστε πολύ σκληρά και πολύ γρήγορα και δεν το βλέπουμε αυτό από άλλους καμιά φορά για διάφορους λόγους. Πριν μπούμε όμως στις λεπτομέρειες και κάνουμε ερωτήσεις στους ομιλητές μας να δώσω τον λόγο στην κυρία Γκράου από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν προφανώς τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσουν οι προσπάθειες μετεγκατάστασης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να σημειωθεί η πρόοδος και ήθελα επίσης να αναφέρω πως η Κομισιόν ενημέρωσε για την ε, αποστολή στις ΕΠΑ ότι είχαμε συναντήσει με Twitter, Facebook και Google για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο Επίτροπος είχε μαζί του και υπουργούς από την Μάλτα και την Εστονία. Και θα έχουμε, είχαμε και την ε, συζήτηση βέβαια των υψηλών αξιωματούχων το καλοκαίρι και σημαντικό ήταν ότι ενημερώθηκε και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στους συναδέλφους. Ε, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ την πρέσβη της Μάρτας για την ε, παρουσίαση. Χαίρομαι ε, γιατί οι αποφάσεις ε, του Συμβουλίου ΔΕΗ ευθυγραμμίζονται ε, με τα θέματα που συζητά το Κοινοβούλιο, αλλά είμαι λίγο απογοητευμένος όσον αφορά δύο θέματα τα οποία θα σας αναφέρω. Στις τελικές αποφάσεις το Συμβούλιο αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνει όσο ε, ε, γίνεται περισσότερη ε, πρόοδος στον φάκελο μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό όμως θα είναι ακόμα Μαλτέζικη Προεδρία και ελπίζω ότι το ένσο θα τελειώσει, το θέμα της ΕΑΣΟ θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο. Ε, γιατί θα πρέπει να λήξει αυτό το θέμα ε, με την υπηρεσία ε, ασύλου. Είμαι λίγο απογοητευμένος με το χρονοδιάγραμμα αυτό. Αυτό σημαίνει και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρωθεί το φάκελος αυτός κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν με ικανοποιεί απολύτως είναι το εξής. Το Συμβούλιο θέλει να δεσμευτούν όλοι για το αιτίας, το, το σύστημα ε, εισόδων-εξόδων. Ε, το Συμβούλιο λέει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου θα πρέπει να ε, υπάρξει συμφωνία και να δεσμευτεί και το, και το Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι η προτεραιότητα για το Συμβούλιο είναι το αιτίας και το σύστημα εισόδων-εξόδων. Ε, αυτό σημαίνει όμως ότι θα αρχίσει να ε, είναι λειτουργικό μετά το 2020. Ωστόσο μέχρι τότε τι γίνεται. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις τώρα. Κατά την άποψή μου θα πρέπει η λύση να βρεθεί εντός των πλαισίων του συστήματος ΣΥΣ. Ε, συζητήσαμε πριν από λίγο τις, προτάσεις της Κομισιόνα. η ΣΥΣ είναι η καλύτερη βάση και πιστεύω ότι αυτό θα, αυτή θα πρέπει να είναι ο που να ακολουθήσει ε, το Συμβούλιο ε, και επομένως όσον αφορά την ασφάλεια θα πρέπει πρώτα το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν να είναι πρώτο και μετά ε, και άμεσα και μετά τα υπόλοιπα. Είμαι λίγο απογοητευμένος λοιπόν γιατί φαίνεται ότι το Συμβούλιο δίνει προτεραιότητα στις δύο άλλες βάσεις δεδομένων και όχι στο ΣΥΣΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Η κυρία Ντάλη θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, πρέσβυρα. Θα ήθελα εγώ να εστιάσω σε δύο διαφορετικές πτυχές. Πρώτον, μετανάστευση. Αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα και είπατε ότι βάρος ε, ρίχνεται κυρίως στην εφαρμογή της διακήρυξης της Μάλτας και πώς μπορούν να συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή και προφανώς η έμφαση που πρέπει να δοθεί ε, στη δουλειά με τους διεθνείς εταίρους. Όμως ε, εμείς ενδιαφερόμαστε στο τι συμβαίνει με τα κράτη-μέλη και μεταξύ κρατών μελών. Και ο Καρμελοντέλα, ο Υπουργός Εσωτερικών στη Μάλτα, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τον τομέα αυτόν, δήλωσε, και δεν ήταν η πρώτη φορά που το είπε, ότι ε, ο χρόνος έχει απόλυτη μεγάλη σημασία. και θα δούμε και άλλες ε, τραγωδίες ε, στην Μεσόγειο, στην κεντρική Μεσόγειο το καλοκαίρι μόλις φτιάξει ο καιρός. Και είναι ήδη τέλος Μαρτίου. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, το συζητάμε εδώ και πολλούς μήνες. Ξέρω πως η Προεδρία της Μάλτας κάνει ό,τι μπορεί. Όμως ε, φαίνεται ότι το Συμβούλιο δεν έχει τόση όρεξη και υπάρχει και αυτό το οποίο είπε ο υπουργό Αμπέλα ότι η εφαρμογή της μετεγκατάστασης ε, είναι μηδενική. Και βεβαίως ε, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Είπατε να αυξηθεί η εφαρμογή, όμως τι εμποδίζει τα κράτη-μέλη από το να εφαρμόσουν αυτά τα οποία έχουν αποφασίσει. Αναφέραμε την Ιταλία και την Ελλάδα και μιλάμε για πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με το πρόβλημα. Πώς ε, το αντιμετωπίζει το Συμβουλίο. Δεν υπάρχει καμία όθηση, δεν υπάρχει όρεξη να κάνουν κάτι. Και ε, πηγαίνει από τον ένα χρόνο στον άλλον. Μια άλλη ερώτηση. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν ε, η απάτη με τα ταξιδιωτικά έγγραφα και το Συμβούλιο εφέτησε συμπεράσματα ενό σχεδίου δράσης για να απαντήσει αυτή την απάτη. Τα συμπεράσματα εστιάζουν στην ανάγκη πιο ασφαλών εγγράφων, ε, μια επανεξέταση της ε, βάσης δεδομένων φάντο και αλλαγή της νομικής βάσης. Ε, και ο συνάδελφος ανέφερε το πώς ε, το πρωί συζητήσαμε το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και το άρθρο 36 το οποίο περιλαμβάνει ελέγχους για τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν τι συζητήσατε στο Συμβούλιο. Είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό το σύστημα και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνουν δύο φορές τα ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο, στον κύριο Ντεπρέ. Ε, ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την ε, ενημέρωση από την Προεδρία του Συμβουλίου και αποκόμισα την εντύπωση ότι το τελευταίο συμβούλιο έγινε σε κλίμα ε, πολύ χαρούμενο έως και εφο, εφορίας ε, κλίμα. Αλλά εγώ από αυτά που διάβασα στον τύπο ε, είναι καταρχήν ότι η Αυστρία ζήτησε να μην υποχρεωθεί να συμμετέχει στη φάση της μετεγκατάστασης που είναι κανονικά υποχρεωτική αρχή για τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο που διάβασα είναι ότι η ομάδα Βεϊσεγκράτ ε, εκπώνησε δικό της ανακοινωθέν τύπου, στο οποίο έλεγε ότι αποκλείεται οι χώρες της ε, ομάδας Βίσεγκρατ ε, να υποκύψουν στον εκβιασμό και στις επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διάβασα στον ανακοινωθέν τύπου της ομάδας των χωρών Βίσεγκρατ. Οπότε ε, δεν ήταν τόσο χα, χαρούμενο το κλίμα ή ουδέτερο όπως το περιγράψατε στην έκθεση που μας κάνατε. Οπότε τι προτείνετε να κάνει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εδώ ενέχεται και το ίδιο το Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή είπε ότι δεν θα διστάσει να εφαρμόσει τις εξουσίες της ε, όπως κατοχυρώνονται από τη συνθήκη. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Επίσης, ε, μια άλλη πληροφορία που με συγκλώνησε είναι ότι η Ουγγρική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει συστηματική κράτηση των ετούντων άσυλο. Αυτό το εξετάσατε καθόλου το Συμβούλιο. Ε, μπήκατε στον κόπο να εξακριβώσετε κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι και θεματοφύλακα των συνθήκων, πρόκειται να αναλάβει δράση στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Ταπρέ. Να προσθέσω κι εγώ μια συμπληρωματική ερώτηση και να κάνω και μια παρατήρηση. Άκουσα και από τις 28 χώρες μέλη ότι φυσικά θα ήθελα να βοηθήσουν τους γνήσιους πρόσφυγες και όχι απλώς τους παράτυπους μετανάστες. Ερωτώ λοιπόν, αν όντως έχουν αυτή την πρόθεση, γιατί δεν ενισχύουν την συνεργασία τους με κάποιες οργανώσεις για να αυξηθεί ο αριθμός των επανεγκαταστάσεων, ώστε να βοηθήσουν τους ε, γνήσιους πρόσφυγες, γιατί νομίζω ότι άλλα τα λόγια τους με τις αγαθές προθέσεις και άλλα αυτά που κάνουν. Σε ό,τι αφορά την κρυπτογράφηση, αυτή τη βδομάδα ακούσαμε και είδαμε κάποια μηνύματα ότι φυσικά χρειαζόμαστε κρυπτογράφηση, και χρειαζόμαστε end-to-end -end ε, κρυπτογράφηση, όχι μόνο για επιχειρήσεις, αλλά και από ιδιώτες. Και θέλουμε να έχουμε και ένα μηχανισμό προστασίας, ε, αλλά να μπορούμε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις να εξετάζουμε τις ανακοινώσεις του Α ή του Β. Δεν είμαι βέβαια εμπειρογνώμονας, αλλά θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχουν καμιά ιδέα πώς μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή να ε, διαβάζουν κρυπτογραφημένες ανακοινώσεις χωρίς να υπάρχει ένα τέτοιο παραθυράκι, να υπάρχει δυνατότητα αυτής της κερκόπορτας. Ε, για το αιτία στο σύστημα πληροφοριών και άδεια ταξιδίου, μία πολύ ε, ε, σύντομη ερώτηση. Από ό,τι ξέρω, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για το σύστημα PNR. Πιστεύετε αν σπεύσουμε με την απόφαση για το ΕΤΙΑΣ ε, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί και στην πράξη το σύστημα. Έχετε κάποια ιδέα ως προς το χρονοδιάγραμμα τα κράτη-μέλη τουλάχιστον. Αυτά και τώρα η πρέσβη Μπονίτσι. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και μετά βεβαίως η Κομισιόν μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, θα απαντήσω πρώτα στο θέμα της πρότασης για το ΕΑΖΟ. Ναι, είπα το συντομότερο δυνατόν, γιατί ελπίζουμε να είναι και πριν τον ε, Ιούνιο. Ε, και δεν θέλω να το προσουζέψω. Έχουμε συνεργασία και με τους ε, βουλευτές, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε. Να τα καταφέρουμε. Επίσης τέθη ένα ζήτημα για την είσοδο, έξοδο και αιτιάς. Όπως είπα, ξεκίνησε ο πολιτικός ε, τριμερής ε, διάλογος. Υπάρχει πολλή πολιτική δουλειά που γίνεται και ελπίζουμε να κλείσει και αυτό όπως μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το τέλος Ιουνίου με το αιτίας ελπίζουμε να έχουμε μια θέση του Συμβουλίου πριν από το τέλος Ιουνίου με το αιτίας όπως ξέρετε είναι πολύ πιο πολύπλοκο οπότε ελπίζουμε να τα καταφέρουμε Παράλληλα βεβαίως δουλεύουμε και για το SIS. Ήταν εδώ πέρα οι δικοί μας ε, το πρωί για να προσπαθήσουν να επιταχύνουν ε, την δουλειά επί του συστήματος γιατί είναι ένα υφιστάμενο σύστημα. Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Πολλά βεβαίω ακόμα πρέπει να απαντηθούν. Αλλά πρέπει να κινηθούμε και γρήγορα με τα μέσα που υπάρχουν ήδη. Συμφωνώ πλήρως. Επίσης, για το θέμα της ε, δήλωσης ε, της Μάλτας. Ε, θα απαντήσω στα Μαλτέζικα. Πολύ δουλειά έχει γίνει πριν από την Σύνοδο Κορυφής στην Μάλτα για να προετοιμάσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Όμως, έχουμε ένα σχέδιο δράσης κάτι το οποίο σημαίνει ότι συναντιόμαστε τακτικά με όλους τους ενδιαφερόμενους και επίσης συναντιόμαστε στο λεγόμενο IPCR και ε, βεβαίως ε, πέρα από όλα τα άλλα και τα κράτη-μέλη και έχουμε και διεθνείς ε, οργανισμούς ε, και ευρωπαϊκές υπηρεσίες που έχουν έναν ρόλο στην ε, εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Όπως ξέρετε η κατάσταση είναι ευαίσθητη γιατί προφανώς εξαρτώμεθα από την Λιβύη. Όμως, πολλή δουλειά γίνεται έργα, τα οποία επίσης εγκρίνονται από την πλευρά της Κομισιόν για να εφαρμοστούν από αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς, Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και η Πατερμοστία του ΟΗΕ. Και είναι πάρα πολύ ε, ισχυρή η εταίρη μας. Προφανώς βεβαίως δεν μπορούμε να βιαστούμε με αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά παρακολουθούμε την εφαρμογή σε τακτική βάση και προχωράμε. Η εκπαίδευση που έπρεπε να γίνει στην Λιβική Ακτοφυλακή έχει γίνει και τώρα περνάμε στα πιο πρακτικά ζητήματα Το σκεφτικό δηλαδή είναι να ε, μπορούν να προστατεύσουν μόνοι τους ε, τις ακτογραμμές μετά. Συνεργαζόμαστε και με τις κοινότητες στην Λιβύη, στην ακτή αλλά και στον νότο της χώρας πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η διακίνηση, η λαθροδιακίνηση έχει γίνει πλέον βιομηχανία ολόκληρη σε τέτοιες χώρες. Οπότε πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις κοινότητες. Να βγάλουν τα προστοζήν με άλλον τρόπο. Αναφέραμε και την μετεγκατάσταση ήταν μια συζήτηση που κάναμε στο γεύμα η Μαλτέζα υπουργό με τον Επίτροπο ζήτησαν αυτά τα κράτη-μέλη να συνεχιστεί η εφαρμογή ε, των ε, κοινών μας αποφάσεων ε, και πρέπει να προχωρήσουμε αλλιώς θα χάσουμε την αξιοπιστία μας εάν παίρνουμε αποφάσεις και δεν τις εφαρμόζουμε παρόλα αυτά ενθαρρυντικό ήταν ότι πολλά κρατημέλη και συνδεδεμένες χώρες επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα εφαρμόσουν τις ε, δεσμεύσεις τους ε, πριν από τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι έχει γίνει κάποια δουλειά. Η διαδικασία είναι δύσκολη. Γιατί δεν είναι όλοι επιλέξιμοι για κατάσταση. Οπότε όταν αποφασιστεί πρέπει να δούμε ποιος θα πάει πού μαζί με τις ε, προσφορές που έχουμε. Οπότε η διαδικασία είναι αργόσυρτη. παρόλα αυτά Έχουμε κάποιες προσφορές ε, και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετεκατασταθούν και ελπίζουμε μέχρι το τέλος ε, Σεπτεμβρίου να μπορούμε να επιτύχουμε πολλούς από τους ε, στόχους που έχουμε. Η κυρία Νταλή επίσης αναφέρθηκε στην απάτη για την ακρίβεια στα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Πράγματι, οι διαδικασίες αυτές είναι χωριστές. Έχουμε δύο προτάσεις χωριστές. Σχετίζονται όμως, όπως σωστά είπατε, και πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να φροντίσουμε να ταιριάζουν οι διαδικασίες και δεν έχουμε επανάληψη. Όπως όλοι ξέρουμε, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Και δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Να σας πω, λέει η Πρόεδρος, ότι ελπίζω οι διερμηνείς μας να μας δώσουν άλλα 10 λεπτά για να συνεχίσουμε την συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είπα. Ναι, θα αφήσω τότε τα τελευταία λεπτά στην Κομισιόν. Είπα όσα είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το ερώτημά σας, ε, κύριε Ντεπρέ, ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να μιλήσουν οι πρόσωποι ε, του, της Γενικής Διεύθυνσης Home, αλλά πρέπει να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξακολουθεί να ελέγχει όλα τα νομοθετήματα και τις αποφάσεις σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα αναφορά τώρα την κρυπτογράφηση ε, στο Συμβούλιο ε, αναφέρθηκε ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έγκαιρο και όχι μόνο από άποψη τεχνολογική αλλά και κυρίως ε, όσον αφορά τις υπόλοιπες διαστάσεις ε, του θέματος. Ε, αυτή τη στιγμή συζητάμε και με την Ουάσιγκτον τα θέματα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας. Από εδώ και στο εξής νομίζω ότι είμαστε σε καλή θέση όσον αφορά τις e-evidence. Έχουμε την τεχνική δυνατότητα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ε, καλά εργαλεία αμοιβαίας αρρωγής και πώς μπορούμε να βρούμε ε, το σωστό νομικό εφαρμόσιμο πλαίσιο. Uh, ε, όσον αφορά την ε, προκρυπτογράφηση, το θέμα δεν έχει οριμάσει ακόμα. Πρέπει να, συζητούμε, να συζητήσουμε ακόμα με τους ε, παρόχους, με τους operators, τους διάφορους φορείς. Στην... Κοιτάξτε, ε, όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα για την κρυπτογράφηση, αν με ρωτάτε αν μέχρι τον Ιούνιο θα μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δεν μπορώ να σας απαντήσω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Θα δούμε. Για τα υπόλοιπα σας παραπέμπω στο συνάδελφο. Πρόεδρος, ε, να επανέλθω στην εκπρόσωπο της DG Home, αν θέλει να μιλήσει. όσον αφορά την κατάσταση. Όντως, ε, περιμένουμε ε, να δούμε πώς θα προχωρήσει η υλοποίηση και βεβαίως εμείς ε, θέλουμε να προχωρήσουμε, να προχωρήσει η διαδικασία, να πιέσουμε ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και θα κάνουμε αξιολόγηση το Σεπτέμβρη. Όσον αφορά το άλλο θέμα για την Ουγγαρία, η Κομισιόν έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την Ουγγρική κυβέρνηση και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν. Ε, συζητούμε τα ζητήματα αυτά με την Ουγγαρία απευθείας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πάντα είναι καλό να έχουμε επιπλέον συζητήσεις. Νομίζω ότι κάπως διέκοψα την κυρία Μπονίτσι, αλλά έχω την αίσθηση ότι απαντήσατε στα περισσότερα, επομένως δεν χρειάζεται να ξαναπάρετε το λόγο. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρίαση να θυμηθείτε εσείς που δεν φεύγετε απευθείας για τα σπίτια σας ότι θα ξαναέχουμε συνεδρίαση στις 2 το απόγευμα στην ίδια αίθουσα.